Good morning everybody. Καλημέρα σας. Θα αρχίσουμε αυτό το εργαστήριο τώρα. Θα μιλήσω σου ειδικά. Λοιπόν, προετοιμαστείτε με τα ακουστικά σας. Ε, Λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σεμινάριο αυτό, στο εργαστήριο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFR, που είναι ένα τμήμα των διαδικασιών που μας απασχολούν. Πρέπει να γνωμοδοτήσουμε από αυτού και θέλουμε το προτέρα να ενημερωθούμε. Θα ακούσετε μία σειρά παρουσιάσεων από εμπειρογνώμονες Και αυτή η έκθεση εδώ μας ε, μεταβιβάζει πληροφορίες, ε, στοιχεία για να μπορέσουμε να δούμε πώς οι οικονομικές πτυχές μπορούν να ενταχθούν στην ζωή. Ε, αυτό λείπει γιατί νομίζω ότι οι οικονομολόγοι ασχολούνται μόνο με αριθμούς και με στατιστικές και ξεχνούν ότι όλα αυτά καλύπτουν ανθρώπινες ζωές και γι' αυτό θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω όλους τους εμπειρογνώμους, το Ίδρυμα Τζάκομου Πρωτοτίνη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Για να εξετάσετε την διάσταση του φίλου στο θέμα αυτό. Τον Αλπέτο Γκόβι επίσης θέλω να χαιρετήσω εγκάρδια το σενάριο αυτό υποδιαιρείται σε μια σειρά τμήματων. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στην κυρία Ζούπερ, την εισηγήτρια της Επιτροπής μας. Μετά θα ακούσουμε έξι μικρές παρουσιάσεις για οικονομική ανεξαρτησία, παιδεία, υγεία, περιβάλλον, μαρία, βασικά δικαιώματα και εξωτερική πολιτική. Μετά από κάθε παρουσίαση μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες, αλλά σύντομες, συγκεκριμένες ερωτήσεις, για να μπορέσουμε να προλάβουμε να έχουμε και τις απαραίτητες απαντήσεις. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα ήθελα να σας καλωσορίσω και καταρχήν να δώσω το λόγο στην κυρία Σούμπερ την εισηγήτρια. Bom dia a todos. Ehm, eu vou falar em português. Ehm, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους προσκεκλημένους, τους συναδέλφους, τους συνεργάτες τους. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είμαι εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή. Μεν, αλλά είναι μια κληρονομιά που πήρα από μια βουλευτή η οποία απεσύρθη το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα, την ε, Χίντα Φιγκερέντο. Θα εργαστώ λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα, κάτω των δυνατόν, προσπαθώντας να παρουσιάσω τις βασικές γραμμές ε, του κειμένου γιατί εδώ πρέπει να γνωμοδοτήσουμε. Και για την προετοιμασία της γνωμοδότησης αυτής είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το εργαστήριο, αυτό το σεμινάριο που έχουμε σήμερα, γιατί πρέπει να ακούσουμε τις απόψεις των πυρογνωμόνων. για να μπορέσουμε τις δικές σας παρουσιάσεις να τις ενσωματέσουμε στο πολιτευσιο δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, ιδίως όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των φύλων. Καταρχήν θα ήθελα να σκιαγραφίσω το θέμα μας. Αυτή τη στιγμή ζούμε μία κρίση μεγάλη και ε, έχει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει στην ισότητα και στην ε, δυνατότητα οι πολίτες να μπορούν να δράσουν. Δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση κατά τη γνώμη μας παρά η επένδυση στην ισότητα των φύλων. Το άρθρο 312 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο να υιοθετείται ομόφωνα υπό τη μορφή κανονισμού του Συμβουλίου. Εκεί καθορίζονται τα διάφορα ποσά και ιδίω τα μέγιστα ποσά ανά κατηγορία δαπανών. Καθορίζονται διάφοροι φάκελοι και πρέπει να εθωρηθούν όλα τα μέτρα ούτως ώστε αυτός ο ετήσιος ε, υπολογισμό να εκτελείται σωστά. Στο άρθρο 8 αναφέρεται το εξή. Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της η Ένωση θα πρέπει να έχει πάντα στόχο την εξάλληψη των ισορροπιών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και πάνω σε αυτό έχουμε συγγνωμοδότηση μια σειρά βασικών σκέψεων. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται μόνο για ένα έγγραφο εργασία. Είναι σαφές κατά μένα ότι η Κομισιόν αναφέρεται στην ανάγκη ευελιξίας και κατά τη χρησιμοποίηση πόρων από το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν ε, αναφέρεται πουθενά ποιο ποσό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ποιο σχέδιο. Παρόλο που θα ήταν σημαντικό κάτι τέτοιο. Για μας πρόκειται για μια σκέψη κλειδί. Υπάρχουν οριζόντιες πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα καθορισμένα ποσά. Υπάρχει η οριζόντια ε, κατεύθυνση οι οριζόντιοι στόχοι, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε συγκεκριμένα για κάθε συγκεκριμένο στόχο με συγκεκριμένο ποσό. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλό να γίνει. Επίσης, το πρόγραμμα Progress θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και πόροι για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτά που προβλέπουμε και στο πρόγραμμα Δάφνη και στο πρόγραμμα Progress που είναι για την ισότητα. Το πολιετές ε, πλαίσιο όμως δεν αντικατοπτρίζει τη σημασία της ισότητας. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα ούτως ώστε οι πόροι που διατίθενται για την ισότητα να μπορούν να χορηγηθούν καταρχήν και χρησιμοποιηθούν κατά δεύτερο. Θα πρέπει δηλαδή εδώ να παίξουν ένα ρόλο οι αιτήσιοι προπολογισμοί ε, που λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τα συγκεκριμένα προβλήματα. Το θέμα της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών είναι πάντα σημαντικό ε, τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής και θα πρέπει να είναι σημαντικό τμήμα της πολιτικής αυτής και γι' αυτό θα πρέπει και συγκεκριμένα να χρηματοδοτηθεί. Ξέρουμε όλοι βέβαια ότι υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης, ακόμα και όσο αναφορά τον Οργανισμό ε, Ισότητας Φύλων. Και θεωρούμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει αναγκαστικά συγκεκριμένες καθευτερές γραμμές για την Κομισιόν θα πρέπει να λεχθεί προς την Κομισιόν ξεκάθαρα ότι θα πρέπει στους ετήσιους προπολογισμού να προβλέπονται συγκεκριμένα ποσά για την χρηματοδότηση της ισότητας και των προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα. Αυτό θα πρέπει πραγματικά κάθε φορά να αποδεικνύεται. Δηλαδή να μην είναι μόνο ευχολογίες αυτά που λέμε για την ισότητα, αλλά να εφαρμοστεί στην πράξη από την Κομισιόν. Κατόπιν δύο λόγια για τις μη κυβερνικές οργανώσεις και τα σχέδιά τους. Ακριβώς σε αυτό το τομέα των δικαιωμάτων γυναικών οι μη κυβερνικές οργανώσεις έχουν πολλά πετύχει. Οργανώσει γυναικών, συνδικάτα κλπ. Και εδώ είναι σημαντικό νομίζω να διαθέσουμε πόρους. Βέβαια, όχι πάντα το ίδιο ποσό, ίσως ε, χαμηλότερα ποσά ή ίσως και υψηλότερα. Ανάλογα. οργανώσεις οι οποίες εργάζονται επί τόπου θα πρέπει να έχουν και μία βασική οικονομική εξασφάλιση αν θέλετε, να έχουν μία βάση απάνω στην οποία μπορούν να στηρίζονται. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μόνο συγκεκριμένα ε, σχέδια ή προγράμματα των μη των οργανώσεων, αλλά να δεδεθούν αρκετοί πόροι, ώστε αυτές οι οργανώσεις να λειτουργούν καθημερινά να χρηματοδοτούμε δηλαδή ένα βασικό δυναμικό εργασία αυτών των ε, οργανώσεων. Και για να ολοκληρώσω, θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί η Κομισιόν επαναλαμβάνει όλα τα ίδια σφάλματα. Δηλαδή μιλάει για εξοικονομήσεις, ορθογωρισμό, περικοπές. Δεν επιτρέπεται όμως να λέμε πάντα τα ίδια και τα ίδια, να πούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε πιο ορθολογικοί, να εξοικονομήσουμε περισσότερο και μετά συγκεκριμένοι στόχοι να μην χρηματοδοτούνται επαρκώς λόγω των πολλαπλών περικοπών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα κατά νου ότι η χρηματοδότηση για την ισότητα δεν θα πρέπει να εξαφανιστεί. Αυτός ο όρος δηλαδή ευελιξία που αναφέρεται από την Κομισιόν ομολογώ ότι με ανησυχεί. Θα πρέπει, και το τονίζω για άλλη μια φορά, να έχουμε συγκεκριμένους στόχους για την ισότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Αναφέρθηκα στην απαραίτητη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, αναφέρθηκα στο πρόγραμμα Δάφνη που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για να εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών. Δεν θα αναφέρω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο, γιατί και εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα σημεία για την ισότητα. Και εδώ θα πρέπει να ελέγχουμε το θέμα το οικονομικό βέβαια. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή που προετοιμάζεται το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί η ισότητα είναι κάτι που είναι σημαντικό και για την εξωτερική εργασία της Ένωσης. Και εκεί προβλέπονται κάποιοι πόροι. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις Διαφάνει ήδη ότι η Κομισιόν δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδης όσον αφορά τον, την κατεύθυνση που παίρνει αυτό το έγγραφο εργασίας. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι στόχοι της ισότητας είναι εξασφαλισμένοι σε ένα πιο γενικό πλαίσιο ήδη. Και αυτό πιστεύει η Κομισιόν ότι προβλέπεται από την ίδια στο πολιετές τη δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς όμως θεωρούμε ότι για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών δεν αρκούν γενικές παρατηρήσεις. Τα γενικά καλά είναι, τα ειδικά είναι πολύ καλύτερα. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Θα σταματήσω εδώ και είμαι σίγουρη ότι αυτό το σεμινάριο σήμερα θα μας δώσει πολύ καλές ιδέες με τις οποίες θα μπορέσω να εμπλουτίσω το έγγραφό μου. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζούμπερ, και περνάμε αμέσω στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την κυρία Μπέτσιο, η οποία θα λάβει το λόγο για μια εισήγηση ως προς τη μέθοδο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου στον προϋπολογισμό. Παρακαλώ. Okay. Hello everybody. Uh... Χαίρετε. Έχω ο καθήκον σήμερα. Έχω πολύ σύντομα καταρχάς να σας παρουσιάσω τη μεθοδολογία πίσω από τις πέντε παρουσιάσεις που θα ακούσετε σε διαφορετικά και ειδικά θέματα. ω αναφέρουμε στη γενικότερη διαδικασία για ενσωμάτωση τη διάθεση των φύλων στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Η ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου στον προπολογισμό είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Η ποιότητα όμω του αποτελέσματο, και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτή την έννοια, ξεκινώντα, εξαρτάται όχι μόνο από την ποιότητα τη ανάλυση, αλλά και από την ποιότητα τη πληροφορία. Το κύριο μήνυμα λοιπόν στις ε, μεθοδολογικές αυτές σημειώσεις είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Είναι όμως και πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σε μέχρι ποιο βαθμό μπορέσαμε να προχωρήσουμε και με τι είδους πληροφορίες στη διάθεσή μας ή τι είδους πόρους που ενδεχομένω αφιερώθηκαν σε αυτή την ανάλυση. Εν γέννη, η ενσωμάτωση της αίσθησης του φίλου στον προπολογισμό συνιστά μια συγκεκριμένη υλοποίηση, εφαρμογή στα χρήματα, σε χρηματικούς όρους, οικονομικούς όρους, της ενσωμάτωσής του φίλου. Και αν το δούμε υπό τους γενικούς του όρους, ε, το σύστημα αυτό, η διάσταση αυτή, ε, απαρτίζεται από τρία βήματα. Καταρχάς πρέπει να προσδοριστούν οι επιθυμητοί ενδεχομένω ε, στόχοι. Δεύτερον, εντοπίζονται Εντοπίστε το πώς ε, είναι αντιληπτή ως προς τα ε, συγκεκριμένα ποσά της πιστώσης που προβλέπει ο προπολογισμό διαπάνω του και τρίτον προσπαθεί κανείς να ε, εκτιμήσει πιθανή πιθανό αντίκτυπο αυτών των ποσών και πιστώσεων για να μπορέσει από την ανάλυση του δεύτερου αυτού βήματος να λάβει κάποιες οδηγίες, κάποιες ενδείξεις για το πού πρέπει να πάει με αυτή την ανάλυση. Αυτά που συνέβη λοιπόν, αυτό που έχουμε κάνει εδώ στην, ε, στο σημείωμά μας είναι πολύ λιγότερο από αυτό που σας περιέγραψα γιατί δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες στη θέση μας. Πλην όμως οι πληροφορίες που θα απορρέουν πιστεύω, ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της δουλειάς που προσφέρει η Επιτροπή των Γυναικών, των Δικαιωμάτων Γυναικών, διασφαλίζει την, το σεβασμό των αρχών για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωσή τους στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και στις τακτικές νομοθετικές διαδικασίες που αφορούν την υλοποίηση και τη λειτουργία των κυρίων προγράμματων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν εντός του πλαισίου αυτού του δημοσιονομικού αυτό που προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε εδώ όλες τις παρουσιάσεις που θα ακούσετε ε, ήταν να εξετάσουμε τα έγγραφα και να δούμε τι ενδείξεις μας δίνουν. Πρώτο βήμα λοιπόν, γενικό πρώτο βήμα της ε, ε, εργασίας αυτής ήταν να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε στόχους ειδικού σας προς το φύλλο ρητούς ή σιωπηρούς στα ε, έγγραφα του προϋπολογισμού και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα ποσά συγκεκριμένα. Πόσα σε χρηματικούς όρους. Και να αξιολογήσουμε κατά πόσον οι πολιτικές που σχεδιάζονται είναι σε θέση να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση προς την ε, ε, τις ε, ανισότητες μεταξύ των φύλων. Αυτό θελήσαμε να κάνουμε. Πρέπει να δούμε βέβαια εάν το καταφέραμε και σε ποιο βαθμό το καταφέραμε. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω, όπως άλλωστε είπα και από την αρχή, ότι όταν ε, η δυσκολία που είχαμε ήταν όταν κοιτάει κανείς τα ποσά, βλέπει ε, Φερρυπίν ε, σε ένα κεφάλαιο ή σε ένα τίτλο ποσά ε, για ένα συγκεκριμένο χώρο και έτσι μπορεί κανείς να δει Φερρυπίν τι ποσό χορηγείται εγγράφεται στον προπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του στόχου της αγοράς εργασίας και τα λοιπά, υπό την έννοια και την προοπτική της ισότητας των φύλων, αλλά δεν βλέπει πουθενά μια συγκεκριμένη διέρεση των ποσών και συγκεκριμένες κατανομές. Άρα αυτό δυσκολεύει πολύ περισσότερο την εκτίμηση του πόσα θα είναι τα πραγματικά το κονδύλια που μπορεί να δαπανηθούν και βέβαια του, απο, αποτελέσματος που μπορεί να επιφέρουν. Ένα άλλο θέμα, στο οποίο νομίζω ότι έχει δυνατότητα άμεση παρέμβαση Επιτροπής, είναι ότι βρίσκονται μέσα στον προπολογισμό κατακαιρματισμένα διάσπαρτα τα στοιχεία που αφορούν προηγούμενη αντίστοιχη μελέτη για τη διάσταση των φύλων. Και έτσι δεν μπορούμε να δούμε εάν υπάρχει κάποια πρόοδος. Καθώς η ευθύνη λοιπόν για τις δαπάνες αυτές ε, να πρόκειται στα κράτη-μέλη, πολλές φορές οι πληροφορίες για, την για τον ε, ε, ουσιαστικό αντίκτυπο των μέτρων δεν είναι διαθέσιμες. Εάν λοιπόν, είναι, αν λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες, δυστυχώς είναι και διάσπαρτες. Και άρα είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τι συγκεκριμένο ποσό ή μέρος ποσού χορηγείται για ποιο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο περιορισμός μας και μέσα στον περιορισμό αυτό, μέσα στα όρια αυτά και μόνο μπορέσαμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας τις πέντε προτάσεις, τα πέντε σημειώματα. Προσπαθούμε λοιπόν να απαντήσουμε στα εξή ερωτήματα. Ποιο θα πρέπει να ωφελείται από, τον, από την παρέμβαση, το στόχο δηλαδή, τι ποσά θα πρέπει να ε, γράφονται και συγκεκριμένα τι είδους ε, επίπτωση, αντίκτυπος προς τα φύλλα από την παρέμβαση αυτή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα. Διότι βλέπουμε ότι εν τέλει μόνο ως προς τα ε, σώματα εξωτερικής δράσης υπάρχει ουσιαστική ε, καταγραφή αυτής της διάστασης ε, στα ποσά δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί ως, προσφέρει ως χορηγός σε τρίτα κράτη. Μόνο εκεί θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ουσιαστική εικόνα και προβλέψεις ε, πιθανής ε, απόδοσης των ε, προσπαθειών και αντικτύπου. Αυτό επειδή, αυτό το οφείλουμε στο γεγονό ότι ο ΟΣΑ ήταν, η ΟΑΣΕ ήταν εκείνη η οποία είχε αναλάβει, η ΟΣΑ ήταν εκείνο ο οποίος αναλάβει τη διαχείριση αυτών των ποσών και εκεί πέρα είναι πολύ πιο σαφής η εικόνα στην διάκριση, στην κατανομή μεταξύ φίλων των συνολικών ποσών που προσφέρουν οι χορηγοί. Και χάρη σε αυτό μπορούμε να έχουμε μια ιδέα του τι είδους αξιολόγηση μπορούμε να αναμένουμε. Ε, αυτή είναι όμως η μόνη περίπτωση. Στις άλλες περιπτώσεις είναι πολύ διάσπαρτες οι πληροφορίες και δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα. Αυτά λοιπόν είναι τα σημεία στα οποία θεωρώ ότι χρειάζεται και μπορεί πιστεύω να αναλυφθεί από πλευρά της Επιτροπής σας δράση. Τα πέντε ενημερωτικά αυτά σημειώματα έχουν και θα τα έχετε δει στο φάκελό σας ως στοιχεία την οικονομική ανεξαρτησία, την κατάρτιση, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το περιβάλλον ως αντικείμενο και η δομή τους ε, είναι αυτή την οποία πρόβλεπα ανέφερα και νωρίτερα ε, ποιος, πόσο και τι, δηλαδή αξιολόγηση ε, αντικτύπου. Πρώτο βήμα λοιπόν, ε, το, η ανάλυση του πλαισίου, το ποιος δηλαδή, μία εκ των προτέρων ανάλυση, η οποία μπορεί πιστεύω να πραγματοποιηθεί σε δημοσιονομικούς όρους, με διαφορετικούς τρόπους, σε μία εκ των προτέρων ανάλυση ε, ουσιαστικά νόημα έχει το να έχουμε μια εικόνα, μια ιδέα των κυρίων διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο αναμενόμενο, στην αναμενόμενη έκβαση συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής. Πριν μπορεί να ρωτήσει κανείς και πάλι επανέρχομαι στο θέμα που με ενδιαφέρει και γνωρίζω καλύτερα την οικονομική ανεξαρτησία στην κατάρτιση. Μπορεί να δώσει κανείς κονδύλια για την κατάρτιση για το παρελθόν, το, το προηγούμενο ποσό, όχι τα μελλοντικά. Μπορεί λοιπόν να γνωρίζει ε, ποια εκ, των προτέρων ποια είναι η αναμενόμενη αξιολόγηση αντικτύπου μια συγκεκριμένη ε, πίστοση ε, στην κατάρτιση με στόχο την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και εδώ αναφέρω την κατάρτιση γιατί στο παρελθόν είχαμε αξιολόγηση τέτοια. Που αποδεικνύεται όμως, απεδείχθη όμως ε, αντιπαραγωγική με ε, διαπίστωση ότι τα ποσά του κοινωνικού ταμείου είναι μάλλον εντείνουν τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και το χάσμα αντί να το καλύπτουν. Και έτσι χρειάστηκε να διορθωθεί η ε, έμφυτη σχεδόν ε, μεροληπτική στάση ως προς την κατανομή των ε, ποσών για την κατάρτιση. Δεν ξέρω σε πόσο βαθμό διορθώθηκε αυτό. Αλλά χρειάζεται τέτοιου είδου διορθώση σε διάφορου τομεί. Το δεύτερο βήμα στην ανάλυση είναι το ποιος Επί τη βάση λοιπόν ε, αναθεώρησης ως προς τους στόχους αναφύλω, έχουμε ένα κατάλογο με στόχους και μετά προσπαθούμε να συγκρίνουμε τα έγγραφα την, ε, με τον κατάλογο για να δούμε εάν η κατανομή των πόρων, των, οικονομικών πόρων είναι αντιστοιχή με τους στόχους που έχουν οριστεί. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα και το τρίτο που ανέφερα νωρίτερα. Μία γενική αξιολόγηση στηριζόμενη στην προηγούμενη προσπάθεια, δηλαδή η σύγκριση του καταλόγου στόχων με τους υλοποιηθέντες στόχους, ε, βάσει των δημοσιονομικών μέσων που εξετάζουμε. Με κύριο στόχο για την ε, προσέγγιση αυτή να ρωτήσουμε ε, σε ποιον αποδίδονται τα κονδύλια, σε ποιον έχουν καταναμηθεί τα κονδύλια, σε ποιο ποσό, φερρυπίν, για ένα συγκεκριμένο ταμείο το οποίο στόχο έχει να προστατεύει από τις δυσκολίες ε, της ε, αλλαγής χώρου εργασίας ε, εργαζόμενους που έχουν πληγεί από το φαινόμενο αυτό λόγω της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι, η... ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εργασίας που χάθηκε πρώτη και κυρίως από τον ανδρικό πληθυσμό στην περίπτωση αυτή. Πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο στόχο έχει να βοηθήσει εργαζόμενους που θα χάσει τη εργασία τους κυρίως σε περίοδο κρίσεως και άρα ίσως να δίνει την προτεραιότητα σε θέσεις για άντρες εργαζομένους ε, χωρίς δηλαδή απαραίτητα να στοχεύει στη στήριξη των γυναικών. Άρα υπάρχουν κάποιοι στόχοι οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την ισορροπία μεταξύ των φύλων στην, στην κατανομή των ποσών. Και σταματώ. Είπα ήδη πολλά για το θέμα αυτό. Προχωρώ στο τρίτο και τελευταίο βήμα που αφορά την, τον αντίκτυπο που περιμένουμε να έχει αυτή η δαπάνη, αυτές οι δαπάνες στο σύνολό τους. Εδώ ακριβώς έχουμε τη, ε, τις περισσότερες επίψεις, όχι γιατί δεν υπάρχει επαρκής ανάληψη, αλλά γιατί δεν διατίθεται επαρκής πληροφορίες. συστηματική και συντονισμένη γνώση ως προς της, ε, τον αντίκτυπο των δαπανών που εγκρίνει το Κοινοβούλιο, κυρίως ως προς το θέμα της ισότητας των φύλων, δεν διαθέτουμε. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους, αν υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια det kan också vara... Okej, Mrs. Klass, please. Ja, danke schön. Ich versuche ja zu... Η κυρία Κλάς, προσπαθώ να μάθω σήμερα και το θέμα του προβολισμού ε, σχετικά με το φύλλο είναι πράγμα που με προβληματίζει. Είπατε, κύριε καθηγητρία, ότι θα πρέπει κανένα πρώτον να καθορίσει τους στόχους. Μπορεί για κάθε στόχο να ορίσουμε κατά πρόσωπο πρόκειται για άνδρε ή για γυναίκες που, στους οποίους στοχεύει το πρόγραμμα. Πρόγραμμα, στα, ε, πρόεδρος, θα συλλέξω όλε τι ερωτήσει, και μετά μπορείτε να απαντήσετε συνολικά. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να θέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα της οικονομικής ανεξαρτησίας και να ευχαριστήσω την ε, καθηγήτρια για την παρουσίασή της. Να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στα συμπεράσματα της εκθέσεώς σας παρατηρούμε ότι τα ποσά τα οποία βρίσκονται λόγω του 2014-2020 για το κοινωνικό ταμείο αυξάνονται κατά 6,6% σχετικά με την προηγούμενη περίοδο. Λέτε όμως ότι αυτή η αύξηση δεν αποτελεί μια ε, σημαντική αύξηση των κονδυλίων που χορηγούνται προς υπέρ της ισότητας των φύλων. Παρατηρούμε ότι παρά την σταθερή απόφαση, την συνεχή αύξηση των ε, χρημάτων στον ε, στο κοινωνικό ταμείο τα χρήματα που χορηγούνται στην ισότητα έχουν ε, ποσοστία μειωθεί. Επίσης πάντα παρακάτω όλες ότι η κατανομή των πόρων γίνεται είναι με τέτοιο τρόπο ώστε ευνοούν περισσότερο τις ε, άνδρες από τις γυναίκες. Λέτε επίσης ότι αυτό θα πρέπει να αντισταθμιστεί ε, προσανατολίζοντα τα ποσά του κοινωνικού ταμείου σε θέματα ισότητας των φύλων και ε, ρωτάω τα εξή. Πρώτον, θεωρείτε πως ε, το να χρησιμοποιηθεί μόνο το κοινωνικό ταμείο θα είναι πιο αποτελεσματικό από ότι, από ότι οι δράσεις ε, σε άλλα μέσα και κάτι ακόμα. Ίσως θα έπρεπε να τεθεί αυτή η, επιτροπή, η ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είμαστε εδώ για να συζητάμε τα, όλα τα ζητήματα και ρωτώ τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν ή μήπως εσείς μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω προς ε, όφελος των ε, δράσεων για την ισότητα των φύλων και διερωτώ με αν θα έπρεπε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, για την παγκοσμιοποίηση, να θέσουμε και εκεί συγκεκριμένου στόχου προ την κατεύθυνση τη όρη των φύλων. Και κάτι ακόμα, απευθύνομαι στου συντάκτες αυτή τη μελέτη, διαρωτώ γιατί δεν υπάρχει κάποιο κομμάτι αφιερωμένο στις δράσεις υπέρ των ισότητων των φύλων και που αφορά στην δικαιοσύνη και ε, σας ευχαριστώ. Επιθυμεί κάποιο άλλο να υποβάλει ερώτηση. Όχι. Α, παρακαλώ. Ναταλή Ντύρς από το New Woman. Είμαστε μια οργάνωση που ε, εδρεύει σε 19 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και έχουμε πολλές χιλιάδες μέλη. Έχουμε ε, επίσης μέλη τα οποία δουλεύουν για την θέματα που αφορούν στις γυναίκες. Διερωτώ αν εάν θα μπορούσαμε να είχαμε πρόσβαση σε κάποια κονδύλια από πλευράς κομισιών, διότι έχουμε ανάγκη από χρηματοδότηση και διότι δουλεύουμε σε προγράμματα για τα παιδιά και τις γυναίκες. Η κυρία Μπετίο θα απαντήσει, αλλά να πω ότι αυτή είναι μόνο η εισαγωγή. Μετά θα περάσουμε στο ζήτημα της οικονομικής ανεξαρτησίας. Είτε ακούστηκε μια σχετική ερώτηση. Παρακαλώ εσείς στο βάθος. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Γκρέισα Τάρτ, είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου των Γυναικών στην Μάλτα, εκπροσωπώ εδώ την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε ό,τι αφορά ένα σημείο της ομιλίας κ. Μπέτιο είπε ότι θα πρέπει να προσέξουμε τα προγράμματα και τα μέτρα να μην δημιουργήσουν περαιτέρω διακρίσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω, πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όταν χρησιμοποιούνται τα κονδύλια π.χ. όταν χρησιμοποιούμε κονδύλια για την, ε, για την εξορρόπηση της ε, ε, του εργασιακού βίου και του βιωτικού βίου, πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να πετύχουμε την επιθυμητή ισορροπία. Επίσης ε, θεωρώ ότι σημασία έχει να μπορέσουμε να εξετάσουμε και τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ε, καταναγκαστική μερική απασχόληση και όχι εθελούσια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπέτιο. Αλλά το θέμα της οικονομικής ανεξαρτησίας ε, θα το απαντήσετε μετά, κατά τη διάρκεια της συνεδριάσης, όχι τώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εγώ προκάλεσα την σύγχυση διότι αναφέρθηκα στην οικονομική ανεξαρτησία ως παράδειγμα προτού να μπω σε λεπτομέρειες. Ναι, πολλές από τις ερωτήσεις ε, τις ε, σημείωσα. και ενδεχόμενα μπορούσα να τις απαντήσω αργότερα όταν θα μπούμε στο θέμα. της οικονομικής ανεξαρτησίας. Η πρώτη ερώτηση ήταν γενικού χαρακτήρα. Αν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε στους στόχους Θα μπορούσα να σας αναφέρω ένα ομό παράδειγμα. Θα μιλήσω αργότερα πάντως λεπτομερέστερα. 75% στόχος για την απασχόληση υπάρχει τώρα. Είναι ένα σαφής στόχος αυτό στο 75%. Παίρνετε απόφαση για να μην υπάρχει διαφοροποίηση, διακρίση μεταξύ άνθρωπων και γυναικών. Μπορεί να είναι καλό ή κακό, εντάξει, δεν ξερουμε με συζήτηση. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμα και αν παραμείνετε στο 75% του του στόχου για το 2020 χρειάζεται να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση γυναικών ξεκινάτε από 57% ενώ για τους άνδρες ξεκινάτε από το 58, 57, 58 για τις γυναίκες 70% για τους άνδρες η διαφορά λοιπόν βλέπετε είναι τεράστια 12-13% μπορείτε αλλά πρέπει και πρέπει επίση να κάνετε διαφοροποίηση όχι στους στόχους αλλά την διαδικασία μέσω της οποίας ε, θα καταλήξετε στον ε, επιθυμητό και αυτό στόχο για τους άνθρωπους και τους γυναίκες. Διαφορετικά η πολιτική σας ε, δεν είναι η ορθή. Δεν είναι ζήτημα ισότητας, είναι ζήτημα αποτελεσματικότητας. Όταν έχετε τόσο μεγάλη διαφορά, 70 με 57-58, βλέπετε ότι το χάσμα είναι τεράστιο τούτου λεχθέντος ας ε, μιλήσουμε για οικονομική ανεξαρτησία μισό λεπτό αν την προς την οθόνη Where the presentation slide It is view Okay. Okay, thank you. Now, um, uh, I mean, let me start from... Να ξεκινήσω από τα βασικά. Αυτό είναι χρήσιμο προκειμένου να μην χανόμαστε. Τι σημαίνει οικονομική ανεξαρτησία. Η οικονομική ανεξαρτησία είναι πολλά πράγματα, αλλά αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι πως καλύπτει την αμοιβόμενη εργασία, αλλά καλύπτει και τη μη αμοιβόμενη εργασία και αυτά είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ε, πολιτικές. Σε μια οικονομία της αγοράς, η οικονομική ανεξαρτησία δεν σημαίνει μόνο οικονομική ελευθερία, διότι φυσικά έχει σημασία να ξέρεις ότι τα χρήματα είναι δικά σου, αλλά είναι και ζήτημα κατανομής ε, των ε, εξουσιών στο πλαίσιο της οικογένειας. Γιατί αυτό, δηλαδή η οικονομική ανεξαρτησία έχει αποκτήσει ε, μεγάλη σημασία για τις γυναίκες τώρα, την εποχή μας. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό για την Ευρώπη γενικότερα, διότι μέσω της οικονομικής ανεξαρτησίας της γυναίκας ελπίζουμε να πετύχουμε τους στόχους ε, που η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οικονομικούς στόχους ε, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η ευημερία. Όλοι γνωρίζουμε πως αν το ποσοστό απασχόλησης ε, των γυναικών δεν ε, επιτευχθεί, τότε υπάρχουν πολύ λιγότερες ε, πιθανότητες για την Ευρώπη να ευημερίσει. Γι' αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερον, υπάρχει κίνδυνος να ε, επιστρέψουμε σε προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή να μειωθεί το βιωτικό μας επίπεδο. Θα υπάρξει λοιπόν οπισθοδρόμηση. Ελπίζω να σας έδωσα μια καλή εικόνα και αυτό συνοπτικά, περιληπτικά σας λέει γιατί η οικονομική ανεξαρτησία παραμένει ένα σημαντικό θέμα σε ό,τι φορά τις γυναίκες. Βλέπετε εδώ στον διαφάνεια Υπάρχουν ε, διάφορες κολόνες, ε, κάθε μια φορά 27 υπάρχει φορά μια χώρα, η τελευταία είναι η Σλοβενία. Τώρα για κάθε χώρα έχουμε τη στήλη που ε, αναφέρει κάθε χώρα και βλέπετε εδώ τα ποσοστά που αφορούν τις ε, γυναίκες και, ε, και τη διαφορά ανάμεσα στο ε, εισόδημα των ανδρών και των γυναικών. Το συνολικό λοιπόν εισόδημα έχει χωριστεί Ας πάρουμε τη Σλοβενία. Βλέπετε λοιπόν βαθύ μπλε κάτω-κάτω στη στήλη. Στη Σλοβενία λοιπόν υπάρχει πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικών που δεν έχουν εισοδήματα. Τώρα το επόμενο μπλε θαλασσί αφορά τις γυναίκες που ε, έχουν, κερδίζουν λιγότερα από τους άντρες. Μετά έχετε το γκρι και αφορά στη ζευγάρια που έχουν ισότιμα εισοδήματα και το κόκκινο είναι το κομμάτι αφορά μάλλον το κομμάτι των ζευγαριών που η γυναίκα κερδίζει περισσότερα και το μαύρο, το πάνω πάνω είναι το κομμάτι που αφορά στην οικογένειες όπου μόνο η γυναίκα έχει εισοδήματα. Όσο ανεβαίνετε προς τα πάνω, ε, φτάνετε στα πεδία όπου οι γυναίκες ε, κερδίζουν περισσότερο. Στο κάτω κομμάτι της στήλη ε, συμβαίνει το αντίστροφο. Λοιπόν, σκοπός αυτού του γραφήματος είναι να δείξουμε τις διαφορές ε, που υπάρχουν ανάμεσα στα οικογενειακά εισοδήματα στα κράτη-μέλη. Αν πάρετε εδώ τη Μάλτα, την πρώτη στήλη, βλέπετε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά γυναίκες που δεν έχουν εισοδήματα. Περίπου 60% σε σύγκριση με τη Σλοβενία, όπου είναι το ποσοστό αυτό χαμηλότερο του 20%. Αυτό που μας δείχνει λοιπόν το γράφημα στην ουσία είναι ότι υπάρχουν τεράστιες διακυμάνσεις ακόμα. Και πώς γίνεται η διαφοροποίηση των ζευγαριών αναφορικά με τα εισοδήματα Βλέπουμε λοιπόν ότι Υπάρχουν ε, πολλά κράτη όπου οι άνδρες έχουν το μεγαλύτερο εισόδημα και άλλα κράτη όπου οι γυναίκες, πολύ λιγότερα φυσικά, ε, έχουν το μεγαλύτερο εισόδημα. Η οικονομική ανεξαρτησία λοιπόν αντιμετωπίσει αυτές τις τρεις διαφορές που υπάρχουν. Και ποιες είναι αυτές οι τρεις διαφορές. Διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης, στην εργασία και στους αμοιβέ. Και τρία αυτά, διαφορές, τα τρία χάσματα συμβάλλουν στο να ε, καταρτιστεί αυτός ο πίνακας που βλέπετε και το γράφημα σας λέει ότι απομένουν ένας μεγάλος δρόμος, μακρύς δρόμος μπροστά μας για να καλύψουμε τις διαφορές. Τώρα για τις λεπτομέρειες τώρα της ε, οικονομικής ανεξαρτησίας. Ε, έχουμε εντοπίσει κάποιους ε, στόχους και μετά ακολουθούν οι ζωτική σημασίας στόχοι που στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με την ε, οικονομική ε, ανάπτυξη όπως η στρατηγική 2020, η ισότητα των φύλων ε, και αφού έχει γίνει λοιπόν αυτό το εγχείρημα προσπαθούμε να δούμε πώς από τους στόχους περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Το τρίτο βήμα ήταν να δούμε τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα για την υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων όπως η στρατηγική 2020 και να παρατηρήσουμε πώς προοικοδοτούνται λοιπόν τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα. Το βασικό είναι το κοινωνικό ταμείο, ένα άλλο είναι το ΕΓΑΦ ε, που σας ανέφερα προηγούμενα για την βοήθεια ε, εργαζομένων που έχουν επηρεαστεί από την ε, παγκοσμιοποίηση και υπάρχουν και άλλα ταμεία, θα τα βρείτε στην παρουσίαση που έχετε αναχείραση. Τώρα, η δυσκολία αυτής, αυτού του εγχειρήματο έγινε το εξή. Θα προσπαθήσω να σας ε, καθοδηγήσω. Τώρα, στόχος ε, αυτού του πίνακα είναι να δείξει πως ε, δύσκολο είναι να εντοπίσουμε τους στόχους και σε ποια προγράμματα έχουν συμπεριληφθεί. Και αυτή η δυσκολία επιδεινώνεται από το ότι η ισότητα των φύλων έχει τύχει mainstreaming, τουλάχιστον έτσι μας λένε, αλλά χωρίς περαιτέρω επεξεργασία σχετικά με το πώς η ισότητα των φύλων γίνεται mainstreamed. Ένα παράδειγμα το έχουμε εδώ και το ανέφερα ήδη. Συγγνώμη, λάθος. δεν ε, λειτουργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες μου το ποντίκι. Λοιπόν, οι στόχοι που έχετε είναι να μειώσετε το χάσμα σε ό,τι φορά την ε, συμμετοχή στην απασχόληση. Το ποσοστό απασχόληση, δηλαδή το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται, επί του συνόλου των γυναικών σε ηλικια εργασια εργασίας είναι 57-58% έτσι εκεί κυμαίνεται και για τους άντρε όπως σας είπα είναι 70% άρα στόχο είναι να περιορίσουμε αυτό το χάσμα ανάμεσα στο 57% και το 70% τώρα η στρατηγική του 2020 όπως ε, έχει διατυπωθεί μπορεί να το πράξει, μπορεί να το πετύχει αυτό εδώ ε, ε, ερωτηματικό διότι η διατύπωση είναι 75% ποσοστό απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες. Εντάξει, μπορεί να είναι, πιο, να είναι εύκολο να πάει οι άντρες από το 70% στο 75%. Αλλά είναι εξίσου εύκολο οι γυναίκες το, το 57-58 να πάνε στο 75% δεδομένων των τεραστίων διαφορών που είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Χρειάζεται περισσότερη, καλύτερη διάρθρωση, δόμηση, αποτελεσματικότητα κλπ. Ένα άλλο παράδειγμα, αν θέλουμε το, το active aging, την ενεργό γύρανση, και ένα στοιχείο για την εργασία των γυναικών είναι ότι το ποσοστό απασχόληση είναι χαμηλό σε προχωρημένη ηλικία. Ένας από τους στόχους λοιπόν είναι να εξετάσετε το πρόβλημα των γυναικών σε μεγάλη ηλικία η στρατηγική 2020 έχετε την ενεργό γύρανση αλλά δεν γίνεται αναφορά στο φύλλο αλλά για λόγους δημογραφικούς ε, ε υγείας κλπ η αντιμετώπιση άνδρα-γυναίκα στην μεγάλη ηλικία δεν είναι η αυτή Αυτά λοιπόν ε, αποτελούν τις δυσκολίες ε, του όλου Λοιπόν, ας δούμε το χρήμα. Εδώ μιλάμε για πολλά χρήματα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ε, στην παρουσίαση, αλλά όχι πολλές. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να υπολογίσουμε πώς ε, θα γίνει η κατανομή στα διάφορα κεφάλια, ε, διάφορους ε, στόχους, υποστόχους κλπ. Τι έχουμε λοιπόν. Καταρχήν τα στοιχεία δείχνουν καλά, διότι ο συνολικός προπολογισμός για το διαθροτικό ταμείο έχει αυξηθεί Ξέχασα να σας πω ότι το Διαθροτικό Ταμείο ε, λαμβάνει το 94% των κονδυλίων. Φυσικά μας ενδιαφέρουν και ίσον σημασία προγράμματα γιατί μπορεί να είναι πιο εστιασμένα. Αλλά τα πολλά χρήματα βρίσκονται στο διαθροτικό ταμείο διότι παίρνει περισσότερο το 90% των συνόλου των κονδυλίων. Εδώ έχουμε αύξηση. Ο υπολογισμός, μάλλον τα στοιχεία τα οποία βλέπετε εδώ, λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, είναι σε πραγματικές τιμές, σε περιπτώσει. Και αναφέρει ότι έχει υπάρξει αύξηση. Ο συνολικός προπολογισμός που αφορά στην ε, οικονομική ανεξαρτησία θα είναι τα 90,7 εκατομμύρια. Ε, ε, δισεκατομμύρια, συγγνώμη. Άρα βλέπετε ότι μιλάμε για πολύ υψηλά ποσά. βλέπετε ότι έχει αυξηθεί κατά 7% συνολικό, ενώ η πολιτική συνοχή έχει αυξηθεί 5,6%. Αυτό είναι καλέ νέα για την ισότητα των φύλων. Και ναι και όχι. Γνωρίζουμε το σύνολο, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το ποσά αυτά κατανέμονται καταλήλως. Και αυτό αφορά εμάς. Εμείς πρέπει να το εξετάσουμε. Εάν ε, κοιτάξουμε στο το παρελθόν και έχουν υπάρξει σχετικές μελέτες, η ειδική προσοχή στο φύλλο μειώθηκε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα κονδύλια που χορηγούνται στον, ε, στα θέματα ισότητας των φίλων, έχουν περιοριστεί στο κοινωνικό ταμείο. Και αυτό συμβαίνει μόλον, συνέβη μόλον ότι τα συνολικά ποσά αυξήθηκαν. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να γίνει στο μέλλον είναι να δεν μειούμε η προσοχή που αποδίδουμε στην ισότητα των φίλων. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει επίσης επιπτώσεις επί της απασχόλησης Χρειάζεται ως εκ τούτου να τονίσουμε πως ε, θα πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές και να παρακολουθούμε τα ποσά και την κατανομή αυτών. Και μια σύντομη παρατήρηση για να καταλήξω Γιατί όλα αυτά έχουν σημασία. Είπαμε ότι είναι πολλά χρήματα διακυβεύονται. Το είδος των δράσεων που έχουν ζωτική σημασία για την οικονομική ανεξαρτησία λόγω της επικουρικότητας βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών. Αυτές, αυτά είναι αρμόδια. Το Ταμείο τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να ε, αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς, ένα, αποτελέσει ένα σύμβολο και να δώσει κάποιες κατευθύνσεις, κάποια καλά παραδείγματα, βέλτιστες πρακτικές. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά είναι σημαντικά. Χρειάζεται επίσης ε, να γνωρίζουμε ότι η απομάκνηση από τους στόχους ε, συμβαίνει όταν ε, παραχωρείται αρμοδιότητες Νομίζω ότι έφτασα στα συμπεράσματα και να αναφέρω κάτι που είπα για την, για την κρίση. Σε περίοδους κρίσης ε, έχει σημασία να τονίζουμε πως η ισότητα των φύλων απαιτείται, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Είναι εντελώς αναχρονιστικό να θεωρούμε ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί πολυτέλεια Και αυτό έχει αναγνωριστεί και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο θέλουμε λοιπόν είναι η κατάλληλη κατανομή των πόρων για το μέλλον. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους βουλευτές καταρχήν και αν υπάρχει χρόνος και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να σχολιάσει. Παρακαλώ. Κύριε Γιανακουδάκη. Να απαντήσω και στις προηγούμενες ερωτήσεις. Ε, ναι, ναι, ε, θα πάρουμε όλες τις ερωτήσεις και μετά θα απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Τις παλιές και αυτές που θα ακούσετε τώρα. Okay, thank you. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω Ε, ένα πρόβλημα που είχα είναι όσον αφορά τα εισοδήματα και λοιπά αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν κάνετε την ανάλυση αυτή λάβατε υπόψη την ηλικία των γυναικών γιατί υπάρχουν ορισμένες φάσεις στην ε, ζωή μιας γυναίκας που δεν ε, κερδίζει χρήματα στα άλλες που κερδίζει πώς το λάβετε υπόψη σας αυτό. Και γιατί χρησιμοποιείτε τόσο πολύ την αναφορά στο φύλλο. Αυτό είναι σημαντικό όταν είναι κανένα νέος και έχει ορισμένα πράγματα στη ζωή του που έχουν επιπτώσεις σε αυτό το ε, στη ζωή του, αλλά όταν περάσει ηλικία 60, ξέρω εγώ, δεν, οι είναι η γυναίκα του ότι βγαίνει κατά κάποιον τρόπο. και ό,τι και να γίνει δεν ξέρω γιατί χρειάζεται αυτή η διάκριση. Η κυρία Σούβερ έχει το λόγο. Μάλιστα, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, ε, κυρία Πενιόλα. θα ήθελα να σας πω ότι με ανησυχεί το γεγονός ότι οι ανησυχίες που υπάρχουν στο δικό μας έγγραφο είναι ακριβώς ανάλογες με τις ανησυχίες και τα προβλήματα που παρουσίασε η εμπειρογνώμων. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μου απαντήσετε στην ερώτησή μου. Θα προσπαθήσω να διατυπώσω κατά δυνατόν σαφώς. Είναι κάτι το περίο, αν θέλετε σε αυτή την εποχή κρίσης αυτό που θέλω να θίξω. Αν δει κανένα πόσες γυναίκες δεν έχουν εισόδημα. Υπάρχουν ενδείξεις γιατί αυτές οι γυναίκες δεν έχουν εισόδημα. Είναι επειδή είναι άντιες αυτή τη στιγμή ή επειδή αποφάσισαν να οργανώσουν την οικογενειακή ζωή κατά τέτοιο τρόπο και να πούνε εντάξει, ο άντρας θα πάει στη δουλειά του και εγώ θα ασχοληθώ με τα παιδιά. Είναι πολιτιστική αυτή η, η απόφαση. Ποιε είναι οι, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών. Πρόεδρος, κάποιος άλλος που θα θέλει το λόγο. Δεν βλέπω. Λοιπόν, θα μπορείτε να μας απαντήσετε ε, και στις προηγούμενες ερωτήσεις της κυρίας Νερισέβα παραδείγματος χάρη. Um, Θα απαντήσω με τη σειρά που υποβλήθηκαν ερωτήσει. Γιατί όλες οι ερωτήσεις αφορούν βέβαια αυτές τις γραφικές παραστάσεις εγώ δεν πρόφτενα να σας εξηγήσω παρά ε, τα, μισά γιατί δεν προλάβαινα. Εδώ είναι οι υπόλοιπε εξηγήσει. Ε, αυτό η γραφική παράσταση αφορά ε, ζευγάρια σε ηλικία που μπορούν να εργαστούν. Υπάρχει δηλαδή ελεγχόμενος ο παράγων ηλικία. Δεν είναι όποιος τυχαίος. Είναι μόνο ζευγάρια σε ηλικία στην οποία μπορούν να εργαστούν. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, Εγώ δεν έχω αναμίξει ε, μαθητές με συνταξιούχους, με εργαζόμενους κλπ. Όχι. Δεύτερο ερώτημα. Είναι πιο ουσιαστικό. Γιατί εξετάσαμε το θέμα της ενεργούς γύρανσης που εξαρτάται από την χώρα μου να προέρχεται κανένας. Γυναίκες στην ηλικία των 50 και 60, αλλά και άντρε όσο πάει και περισσότερο. Ασχολούνται κατά κύριο ποσοστό σε πολλές χώρες, όχι με παιδιά πια, αλλά με ηλικιωμένους. Λοιπόν, θα πρέπει κανένας να ρωτηθεί τι γίνεται σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα όταν το δει αυτό. Γιατί απορροφά κανένας πόρους ε, για την φροντίδα ηλικιωμένων. Επίσημα ή ανεπίσημα δεν έχει σημασία. Γίνεται. Είναι καλό αυτό μεν, αλλά απαιτεί, πώς να σας το εγρά περιγράψω, απαιτεί κάποια προγράμματα φροντίδας. Εάν ζητάει δηλαδή κανένα από περισσότερες γυναίκες στις χώρες αυτές να εργάζονται εκτός οικογένειας, χρειάζεται ταυτόχρονα να υπάρχουν προγράμματα που θα φροντίζουν τους ηλικιωμένους. Δηλαδή μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι θέμα απασχόλησης πάλι. Ναι, ναι, αλλά ε, είναι και ένα τμήμα της ε, οικονομικής ανεξαρτησίας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πώς σχετίζεται η απασχόληση με την φροντίδα. Δεν μπορεί κανένας να αποχωρήσει τα μένα από τα δε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό το πρόβλημα της ε, ε εργασίας η οποία μισθή δίνεται για τους ηλικιωμένους κατόπιν. Ναι, υπάρχουν ανησυχίε, σωστά, υπάρχουν, αλλά ε, δεν ε, είναι ακόμα καθορισμένα τα ποσά, τα οποία αυξάνονται. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω εδώ κάποια αισιοδοξία ε, και όχι απεσιοδοξία. Όσον αφορά το θέμα του πίνακα οι περισσότερες από τις γυναίκες που δεν εργάζονται είναι οι γυναίκες όχι που είναι άνεργες αλλά που αποφάσισαν ή υποχρεώθηκαν να αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να εργαστούν. Και υπάρχει μόνο ένας άντρας ο οποίος κερδίζει τα χρήματα γυναικών είναι αυτή. Στην ε, γραφική παράσταση δεν υπάρχει όμως διάκριση μεταξύ των δύο. Αν κανένα έχει κάνει την επιλογή αυτή ή αν δεν εργάζεται επειδή είναι άνεργο. Θα πρέπει να έχει κανένα έναν ξεχωριστό βέβαια πίνακα, είναι αλήθεια. Ενώνει δηλαδή αυτή η γραφή παράσταση στις δύο υποθέσεις αυτές. Την ε, ανεργία και την εθελοντική μη εργασία, το πούμε έτσι κατόπιν. Εγώ προσπάθησα να απαντήσω στα ερωτήματα για την διαφοροποίηση των στόχων και ελπίζω να ήμουν επιτυχής. Όταν παρουσίασα τους στόχους για την ισότητα των φίλων και είπα πόσο δύσκολο είναι από την άλλη μεριά να πάρει κανένας αυτούς τους στόχους και να τους ενσωματώσει στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, που είναι πολύ γενικά διατυπωμένη. Λοιπόν, ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας αυτή, ότι είναι σωστό να έχουμε στόχους, ένα φύλλο ή τουλάχιστον μια διαδικασία που μας επιτρέπει να στοχεύσουμε προς την ίδια κατεύθυνση αλλά στοχεύοντας χωριστά τους άντρες και τις γυναίκες. Μετά, έχω εδώ, ίσως παρανοήσει κάτι θέμα για το ταμείο, γιατί συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στο κοινωνικό ταμείο. Αυτό ήταν ή δεν κατάλαβα εγώ, δεν σημείωσα σωστά τα πράγματα. Κοιτάξτε, 94% του προπολογισμού για την οικονομική ανεξαρτησία είναι αυτό. Αν ξεραστεί κανένα άλλος ε, στόχους, ίσως κάποια άλλα ταμεία να είναι πιο ε, κατάλληλα και ίσως μπορεί κανένας καλύτερα να ασκήσει πίεση για αυτά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν θέλουμε να γίνει κάτι πολύ σημαντικό θα χρηματοδοτεί από το κοινωνικό ταμείο. Δεν έχω άλλες ε, καθαρές σημειώσεις εδώ. Αν είχατε και κάποια άλλη ερώτηση παρακαλώ να την επαναδιατυπώσετε και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Okay, we take one, one more question here. Μία, ακόμα, μία ακόμα ερώτηση μόνο, παρακαλώ. Από το Βρυκό Ινστιτούτο για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Έχω μία ερώτηση που, επειδή εδώ στοχεύουμε πολύ στο Κοινωνικό Ταμείο, έχετε λάβει πώς την ανάλυση σα, Έχω δίκιο που το θεωρώ ότι μέσα στα ποσά για το κοινωνικό ταμείο υπάρχουν και κάποια κριτήρια για την ισότητα των ε, φύλων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Παραδείγματος στη Φλάνδρα ξέρω ότι όταν ζητάνε κάποια χρηματοδότηση για κάποια σχέδια υπάρχουν κριτήρια πριν δοθούν τα χρήματα αυτά πρέπει να απαντήσουν σε κάποια ερωτηματολόγια και υπήρχε και ένα σχέδιο όπου υπήρχε ένας σύμφυλος που έκανε ένα σεμινάριο για όλους τους ε, εκείνους που είχαν υποβάλει τα σχέδια αυτά και έπρεπε κανένα να το ξαναγράψει το σχέδιό του για να λάβει υπόψη καλύτερα την ε, διάσταση του φύλου. Αυτά όλα έχουν ληφθεί υπόψη στη δική σας ανάλυση. Και είναι αυτό μια συγκεκριμένη ε, υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή είναι κάτι που ειδικό που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Φλάνδρα. και η ισότητα των φίλων πραγματικά ενσωματώνεται σε αυτούς τους διάφορους στόχους. Αυτό το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μήπως θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να, ε, να κάνουμε αυτό το κριτήριο πιο ισχυρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ που φανταζόσατε ότι θα μπορούσαμε να πάμε σε τόσες λεπτομέρειες. Δεν μπορούσαμε. Αλλά ελπίζω να μπορούσα να σας απαντήσω. Είναι απόλυτα σωστό ότι υπάρχουν στόχοι ανάλογα με το φύλλο, ορισμένοι συγκεκριμένοι, ρητοί και άλλοι ε, πιο ασαφείς για τη στρατηγική του 2020, διότι απλούστατα όλοι ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σημαντική συμμετοχή για να μπορέσουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη. Κάτι υπάρχει λοιπόν εκεί. Επίσης, υπήρχε και ένα θέμα της κατανομής εργασίας μεταξύ στρατηγικής του 2020 και στρατηγικής για ισότητα, όπου εννοείται ότι οι σαφείς στόχοι για την ισότητα που υπάρχουν στη σχετική στρατηγική θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην πολιτική της Ένωσης του 2020. Και περνάω εδώ στο στόχο αυτό, αυτού που κάνουμε. Δηλαδή, χρειάστηκε να δούμε κατά πόσον τα χρήματα αυτά δίνονται στους στόχους οι οποίοι ακόμα και αν συγκεκριμένα λένε ότι είναι για γυναίκες είναι σημαντικά για την ισότητα των φίλων Και το δεύτερο, η διαδικασία που οδηγεί στην δαπάνη ποια είναι και ο έλεγχος των επιπτώσεων των ποσών αυτών είναι σωστά καθορισμένη από σκοπιάς ισότητας φύλων. Πρώτον, δεν μπορούσαμε να περάσουμε στο δεύτερο στέδιο. Και το τρίτο εξαρτάται πολλές φορές από κάθε χώρα. Παρόλο που ίσως υπάρχουν γενικές οδηγίες, κατευθύνσεις γραμμές κλπ. Η συγκεκριμένη εφαρμογή διαφέρει ίσως από χώρα σε χώρα. Και γι' αυτό επέμεινα στην εποπτεία που είναι τόσο σημαντική. Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το πολύ καλό παράδειγμα της Φλάνδρας. Ελπίζω να μπορεί να το ακολουθήσουν και άλλες χώρες. <clears throat> Αλλά δυστυχώ υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο σε άλλον ένα, αλλά πραγματικά ο τελευταίος, τελευταίος, τελευταίος που θα του δώσω το λόγο, γιατί αρχίζουμε να έχουμε καθυστέρηση. Η κυρία Τάτα έχει το λόγο. Παρακαλώ πολύ σύντομη στην ερώτηση και πολύ σύντομη στην απάντηση επίσης. Ευχαριστώ. Ε, ξέρετε όλοι ότι η Κομισιόν προετοιμάζει μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών Διαθωτικών Ταμείων. Διαφορετικά ομοδοποιημένα τα διάφορα προγράμματα, με την ανάγκη να υπάρχει κοινωνική καινοτομία, ε, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εμείς ανησυχούμε στην Επιτροπή μας γιατί δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο και όσον αφορά από πλευρά φίλου. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Δεν μπορώ παρά να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Α, πραγματικά ήταν σύντομη αυτή η απάντηση. Ε, με εντυπωσιάσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπέτιο για την παρουσίασή σας και περνάμε τώρα στην επόμενο σημείο. Θα ήθελα να καλωσορίσω την επόμενη μιλήτρια, την κυρία Μιούλτερ, που θα κάνει μια παρουσίαση 15 λεπτών των αποτελεσμάτων της για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Ένα τέταρτο έχει παρακαλώ. Euh, Θα μιλήσω γαλλικά παρότι οι διαφάνειές μου είναι στα αγγλικά γραμμένες. Θα σας ε, παρουσιάσω το θέμα που έχει να κάνει με την εκπαίδευση και κατάρτιση με εφαρμογή στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα της μεθοδολογίας που σας παρουσίασε νωρίτερα κυρία Μέτσιο. Προσπαθούμε δηλαδή να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι που μπορούμε να διαγράψουμε στο θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με αναφορά στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, να διαγνώσουμε μέσα στα προγράμματα, από τα προγράμματα ποια έχουν να κάνουν με εκπαίδευση και κατάρτιση και ως εκ τούτου σε ποιο βαθμό δίνεται απάντηση στους στόχους αυτούς από συγκεκριμένα προγράμματα που προτείνονται και ταυτόχρονα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε μεταξύ των ποσών που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό ποια είναι τα καταλληλότερα για να τα ανταποκριθούν στους στόχους που ε, έχουν εντοπιστεί. Εκπαίδευση κατάρτιση λοιπόν είναι ένα τομέα ιδιαίτερο στο βαθμό όπου τα άρθρα 165-166 της Συνθήκης Λισαβόνας, στον τίτλο 12 «Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, νεολαία, αθλητισμός» προσδιορίζουν επακριβώς τα όρια δυνατότητας δράσης των θεσμικών οργάνων σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Αρμόδια δηλαδή για τον ε, σχεδιασμό της πολιτικής τους για το περιεχόμενο της εθνικής ε, παιδείας, ε, την περιγραφή του συστήματος, είναι τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποια όρια δηλαδή στις δυνατότητες δράσης. Πλην όμως τα άρθρα αυτά της Συνθήκης του Σαφώνας προσδιορίζουν ξεκάθαρα ότι στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και της επαγγελματικής κατάρτισης στηρίζει, υπάρχει δράση υποστήριξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σεβασμό της αρχής επικουρικότητας και η Ευρώπη διευκολύνει πάντως την επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με την ένταξη και επανένταξη στον χώρο εργασίας. Ο σύνδεσμος λοιπόν μεταξύ της ενημέρωσης και της αγοράς, ε, της εκπαίδευσης καλύτερα και της αγοράς εργασίας ε, πάντοτε ήταν στο επίκεντρο της Ευρώπης, δηλαδή θεωρούταν πάντα ότι η εκπαίδευση είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση, η διατήρηση ενός ανθρώπου, η επανένταξη ενός ανθρώπου στο χώρο εργασίας. Έτσι αντιμετωπίστηκε η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιμετωπίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η στρατηγική της Λισαβόνας του 2000 που είχε σαν στόχο η Ευρώπη να μετατραπεί σε κοινωνία γνώσεων, σε θέματα προηγουμένης, σε, σε τομείς εχμής. και άρα ιδιαίτερη έμφαση στην ε, εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς εχμής για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, σημειώνει μια συγκεκριμένη βούληση για παρέμβαση στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά όπως είπα συμπληρωματικά και ε, με σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Άρα, στα νέα αυτά προγράμματα η εκπαίδευση συνιστά ακόμη μέσων ένταξης ή επανένταξης στον χώρο εργασίας και παραμένει από ό,τι διαπιστώνουμε η ε, εκπαίδευση τρόπος να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Όταν διαπιστώνουμε, όταν κοιτάμε τα δεδομένα της Eurostat, παράδειγμα, με τα ποσοστά της εκπαίδευσης, ασφαλώς και αναμφίβολα, όσο πιο πολλές γυναίκες ε, έχουν, ε, όσο πιο καλή εκπαίδευση έχουν οι γυναίκες, τόσο πιο πολλές είναι και οι πιθανότητες τους να βρουν μια θέση εργασίας. Άρα ο στόχος της αύξησης της απασχόλησης, των ποσοστών απασχόλησης μέχρι το 75% προφανώς και εξυπηρετείται με τη δυνατότητα αυτή της αύξησης δηλαδή του επίπεδου της εκπαίδευσης. Τα μέσα που εξετάσαμε. Ας δω τη γαλλική έκφραση. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. που βλέπετε εδώ στην παρουσίασή μας ως Education and Training 2020. Το πρώτο πράγμα στο έγγραφο αυτό, που είναι και λίγο ανησυχητικό για την ε, δική μας μελέτη, είναι ότι δεν γίνεται ζήτημα, δεν υπάρχει δηλαδή δική ερώτηση ως προς τα φύλλα διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκτός από μια πρώτη ερώτηση, μια πρώτη παρατήρηση που αναφέρει ότι στην αρχή αρχή του κειμένου ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει ισότητα μεταξύ των φίλων στον ε, τομέα αυτό. Αλλά στα συγκεκριμένα προγράμματα δεν υπάρχει άλλη αναφορά ε, συγκεκριμένη. Και αυτό ακριβώς είναι και αξιοσημείωτο και ενσχετικό. Από την άλλη, σημαντικά έγγραφα, σημαντικά νομοθετήματα ευρωπαϊκά ε, που αφορούν είτε προηγούμενες πολιτικές όπως ε, το φύλλο πορείας ε, για το ρόλο των γυναικών 2006-2010, η στρατηγική για την ισότητα 2010-2015, το έγγραφο που θέλει να δώσει μια νέα όθηση στην επαγγελματική κατάρτιση και την ε, επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη με την Ευρώπη του 2020 και το σχετικό προϋπολογισμό ε, αναφέρονται στο πρόβλημα της ε, ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά το πρώτο έγγραφο που είναι σημαντικό, διότι είναι το κατεξοχήν ε, πρόγραμμα για το 2020, δεν καταγράφει αυτή τη διάσταση συγκεκριμένα. Πρώτο λοιπόν, ε, για να καταλήξουμε σε διαπιστώσεις, εάν προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα ως προς την κατάσταση για τα 27 κράτη-μέλη από κοινού, θα ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε κοινά σημεία γιατί η κατάσταση που επικρατεί στα κράτη είναι πολύ διαφορετική. Το να καταμετρήσουμε δηλαδή τι ανισότητε μεταξύ ανδρών και γυναικών στα συστήματα εκπαίδευση και κατάρτιση ανά την Ευρώπη είναι κάτι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλέ ε, ε, ακραίες θέσεις, πολλές μεγάλες διαφορές δηλαδή από τη μία στην άλλη ακραία θέση μεταξύ κρατών και όσο θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Πλην όμως από μελέτες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από άλλες πηγές μπορούμε να εντοπίσουμε έξι τομείς στους οποίους μπορούμε να επισημάνουμε σημαντικές αποκλήσεις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και βέβαια βάσει αυτών των διαφορών προσδορίζουμε και τους έξι στόχους που εντοπίζονται και στη συνέχεια συγκρίνονται με τα, όσα προβλέπουν τα προγράμματα και οι προπολογισμοί. Πρώτον λοιπόν, το πρώτο σημείο έχει να κάνει με τις βασικές γνώσεις μεταξύ κοριτσιών και αγοριών από την στοιχειώδη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και εδώ οι μελέτες PISA του ΩΣΑ επισημαίνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον ως προς την απόκληση μεταξύ ανδρών και γυναικών ή εν προκειμένου κοριτσιών και αγοριών. Αποδεικνύεται, λοιπόν, καταδεικνύεται μάλλον μια σημαντική διαφορά υπέρ των κοριτσιών στο χώρο της ανάγνωσης. Το χάσμα ανοίγει, η ψαλίδα ανοίγει 39 μονάδες κατά μέσο όρο στην Ευρώπη με σημαντικές διακυμάνσεις ε, μεταξύ των διαφορών κρατών αλλά έχουν πολύ σημαντικό πλεονέκτημα τα κορίτσια στην ανάγνωση και την κατανόηση και μάλιστα με αυξανόμενη τάση αυξητική τάση. Ενώ από την άλλη έχουν ελαφρά υστέρηση ή μειονέκτημα ελαφρώ στα μαθηματικά, το οποίο όμως μειονέκτημα είναι ίσον σε σχέση με τη μεγάλη διαφορά που χωρίζει τα κορίτσια από τα αγόρια στην ανάγνωση και την κατανόηση και εν τέλει είναι λίγο πολύ ισότιμες οι επιδόσεις στα, ε, στις επιστήμες. Πρώτο λοιπόν σημείο αυτό και διαπιστώνουμε με την πρώτη ερώτηση που μας απασχολεί, εάν ε, αναλαμβάνονται δράσεις στον τομέα αυτών και εάν υπάρχουν προϋπολογισμοί ε, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Η δεύτερη πρόταση, το δεύτερο σημείο, έχει να κάνει με την ε, έξοδο από το σχολικό σύστημα, την εγκατάλειψη των σπουδών, που πάλι παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των ε, κρατών αλλά και με ποσοστά σημαντικά νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο και, και πάλι σε μειονεκτικότερη θέση βρίσκονται τα αγόρια. Η διακοπή ε, των, σπουδών δηλαδή αφορά περισσότερο τα αγόρια παρά τα αγόρια στις περισσότερες χώρες. Το τρίτο σημείο, γενική εκπαίδευση. Εδώ προφανώς υπάρχει βούληση για αύξηση του επίπεδου της γενικής εκπαίδευσης. Για δε τις διαφορές μεταξύ ανδρών, ε, κοριτσιών και αγοριών ε, που διαπιστώνονται έχουν να κάνουν περισσότερο με τους προσανατολισμούς, δηλαδή μια οριζόντια, ένας οριζόντιος διαχωρισμός στα αντικείμενα σπουδών και στους κλάδους σπουδών. Πιο πολύ δηλαδή τα αγόρια τα βρίσκουμε στην επαγγελματική κατάρτιση που να τους δώσει ε, προσόντα επαγγελματικά νωρίτερα, ενώ τα κορίτσια θα παραμείνουν περισσότερο στη γενική εκπαίδευση. Το επόμενο σημείο αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, όπου βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Τα κορίτσια πάντα, παντού είναι πιο πολύ άριθμα από τα αγόρια, φοιτήτριες πέστος από τους φοιτητές. 55% είναι τα κορίτσια στην ε, ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη και πιο ε, πολυάριθμες επίσης αν κοιτάξουμε τα στοιχεία των πτυχιούχων. Πάλι λοιπόν σε μειονεκτική θέση οι άντρες. Και τα ποσοστά αυτά πάλι αυξάνονται. Η διαφορά αυτή αυξάνεται και ως εκ τούτου γίνεται όλο και πιο σημαντική. Άρα χρειάζεται η προσοχή στο φαινόμενο αυτό. Στο πέμπτο σημείο. Κοιτάμε σε, ποια, σε ποιους τομείς σπουδών έχουν εγγραφεί και εξειδικεύονται οι φοιτητές. Εδώ πάλι βλέπουμε ότι δεν ακολουθούν τους ίδιους κλάδους σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κορίτσια και αγόρια. Οι γυναίκες δηλαδή έχουν μόνο συμμετοχή κατά 30% περίπου και ανάλογα βέβαια με την κάθε χώρα υπάρχουν και αποκλήσεις στα θέματα, στους τομείς της ε, μηχανικής, μηχανολογίας, μαθηματικών, τεχνικών ε, σπουδών εν γέννη. Είναι ε, αυτοί οι μόνοι τομεί στου οποίου δεν είναι πιο πολύ άριθμε οι γυναίκες από τους άντρε, στους υπόλοιπου είναι πιο πολύ αυτό ήταν το πέμπτο λοιπόν σημείο και στόχος ταυτόχρονα. Και στο έκτο έχουμε τις ανισότητες ως προς τη συμμετοχή στην διαβίου μάθηση. Και εδώ πάλι κατά αντίθεση οι γυναίκες έχουν λιγότερη συμμετοχή στην ε, διαβίου μάθηση από ότι οι άντρες. Έτσι λοιπόν προσδορίζουμε με βάση την ανάλυση αυτή τους ε, στόχους στην αριστερή στήλη και με τη μέθοδο που έχουμε προσδιορίσει προσπαθούμε να δούμε εάν στα ευρωπαϊκά έγγραφα ε, νομοθετήματα λαμβάνονται υπόψη αυτή οι στόχοι, αυτές οι ελλείψεις και αυτή οι στόχοι. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο πρώτος στόχος που θα ήταν η εξάλληψη των διαφορών στις, ε, στη βασική εκπαίδευση, στις βασικές γνώσεις δεν λαμβάνεται υπόψη από τη στρατηγική. Μετά έχουμε όμως στόχους που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόορης εγκατάλειψης των σπουδών στα περισσότερα από τα ε, έγγραφα που εξετάσαμε, αλλά κατά τρόπο ουδέτερος προς τα ε, φύλλα για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 που στοχεύει σε μείωση στο 10% των νέων που αφήνουν το σχολείο χωρίς να πάρουν το απολυτήριό τους. Δεν ξεχωρίζει όμως κορίτσια ή αγόρια. Στη στρατηγική για την ισότητα προσδορίστε το φύλλο αλλά χωρίς στόχο ποσοτικό. Άρα ως στοιχείο υπογραμμίζεται αλλά χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Ε, σε σχέση με τα φύλλα, στην ε, ε εκπαίδευση κατάρτιση 2020 στην τρίτη στήλη. Επίση, συμμετοχή των γυναικών στην επαγγελματική κατάρτιση ε, πάλι έχουμε ουδέτερη στάση ω προ τα φύλλα με συγκεκριμένο στόχο στρατηγική 2020 και στρατηγική ισότητα Στρατηγική 2020 έχουμε 40% για τον, για τον πληθυσμό συνολικά των 30-33 ετών για το 2020 με επαγγελματική κατάρτιση η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε ορισμένους τομείς αναφέρεται στη στρατηγική για την ισότητα χωρίς όμως συγκεκριμένο στόχο ποσοτικό και το ίδιο αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη διαβίου μάθηση. Άρα, ορισμένα έγγραφα το, το αναφέρουν, χωρίς όμως συγκεκριμένου στόχους και αυτό ε, συνάδει και με τα σχόλια που έγιναν νωρίτερα για το 75% στην απασχόληση, συγκεκριμένοι στόχοι. Τα δύο προγράμματα που αφορούν περισσότερο την εγκατάρτιση, την εκπαίδευση είναι το Έρασμους που αφορά τους πάντες και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρώτο λοιπόν που έχουμε να πούμε, γιατί βλέπω ότι περνάει ο χρόνος και επιταχύνω, στο πρόγραμμα έρασμου για όλους, Erasmus for All, με προϋπολογισμό 19 δις διαπιστώνουμε με μια ανάγνωση του προγράμματος όπως έχει αυτή τη στιγμή γιατί μπορεί βέβαια να βελτιωθεί ε, ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε φύλλο, δεν υπάρχει καμία ειδική στρατηγική είτε για άντρες είτε για γυναίκες, δεν υπάρχει ειδική πίστοση ε, ως προς τα φύλλα, ούτε συγκεκριμένη δράση ε, του προϋπολογισμού για ε, κάποιες προσπάθειες ε, υπέρ της ισότητας ή στη σχέση με τα φύλλα. Ούτε καν αναφέρεται διατύπωση δεδομένων ειδικών ω προ το φύλλο για να μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια τη μελέτη και την αξιολόγηση. Αντίθετα όμω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που το αναφέραμε και νωρίτερα σημειώνει με ιδιαίτερη έμφαση τη διαφορά του φύλλου και ορίζει προγράμματα με συγκεκριμένους στόχους φύλο ή δράσεις συγκεκριμένα που θεσπίζονται για να, ε, με στόχο να εξαλείψουν τις διαφορές. Ο πίνακας απλώς επιβεβαιώνει αυτή η διαπίστωση που βλέπετε εδώ, δηλαδή ορίζουμε, καταγράφουμε αριστερά τους έξι στόχους στην αριστερή στήλη. Μετά βλέπουμε ότι στον έρασμο, έρασμος για όλους, ε, όλες οι απαντήσεις ως προς τους στόχους είναι αρνητικές, δεν αναφέρεται πουθενά κάτι λεπτομέρες ως προς τα ε, προγράμματα, αν και θα έπρεπε πρώτα να μιλήσω για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, γιατί για αυτά δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά τεκμηρίωση. Τα πάντα δηλαδή θα μπορούσαν ε, να προκύψουν εάν λάβουμε πιο πολλά στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει όμως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαπιστώνουμε ότι για το σύνολο του Ταμείου τα 25 δις μπορεί να έχουν να κάνουν το της εκπαίδευσης και κατάρτισης και πάλι όμως χωρίς να μπορέσουμε να ε, κατακαιρματίσουμε το ποσό αυτό και να, να εντοπίσουμε συγκεκριμένες δράσεις ε, για κάθε φύλλο. Και πάλι οι τομείς και οι στόχοι που έχουμε εντοπίσει δεν λαμβάνονται υπόψη. Και για να κλείσω, και θέλω απλώς να υπογραμμίσω το εξής, ότι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο φαίνεται αυτή τη στιγμή να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα του φύλου και θα μπορούσε ενδεχομένως να φέρει αποτελέσματα ε, σε σχέση με κάποιους από τους στόχους, όχι όλους όμως τους στόχους που έχουν εντοπιστεί, γιατί κάποιοι από τους στόχους δεν λαμβάνονται υπόψη στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Στο Erasmus for All δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα, πολλά μένουν ακόμα να γίνουν, αλλά βέβαια μπορεί και να γίνουν τα πάντα, γιατί είμαστε στην αρχή της ε, κατάρτισης, στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης πάντα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική δυσκολία όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική του gender budgeting, της εγγραφής του προπολογισμού, της διάστασης του φύλου. Γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ και στο συγγνώμη που σας ευχαριστώ, κυρία Μέλτερς. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε ερωτήσεις. Ιάνσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Μόλτερς για την παρουσίαση αυτή για την εκπαίδευση. Ε, έχω υπόβαθρο εκπαιδευτεί στην ε, κατάρτιση ενηλίκων και έχω ασχοληθεί και με θέματα της εκπαίδευσης υπό, ε, υπό το πρίσμα της, κατάρτιση κατάρτισης ενηλίκων πάλι. Όταν λοιπόν συζητούμε την εγγραφή στον προπολογισμό Πρόβλημα είναι βέβαια οι αρμοδιότητες, γιατί η εκπαίδευση, όπως είπατε, δεν, είναι δεν, ανήκουν... Ε, δεν ανήκει σε αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των κρατών μελών και μάλιστα πολλέ φορές και στο τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Είπατε ότι σε κάποια από τα μεγάλα αυτά ταμεία, Εράσμους, ε, Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου και σε άλλα προγράμματα υπάρχει η διάσταση της εκπαίδευσης κατάρτισης. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μπορούμε ε, να κάνουμε μια προσπάθεια και να αλλάξουμε μακροπρόθεσμα τις ε, τάσεις. Ε, θα ρωτούσα λοιπόν το εξής. Σε ποιον τομέα του προϋπολογισμού πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση που θα έπρεπε ιδιαίτερα να παρακολουθούμε τα θέματα της κατάρτισης όπως το Εράσμος, το Κοινωνικό Ταμείο, Περιφερειακή Ανάπτυξη, σε ποιο θα δίνατε πιο πολύ σημασία. Για το τομέα της εκπαίδευσης. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω εάν η εγγραφή των θεμάτων του φίλου, της των φίλων στον προϋπολογισμό καταγράφεται ε, σε εβδομαδιαία βάση και πώς. Ευχαριστώ. Κοίταξα τα διάφορα σημεία από 1 ως 6 και φαίνεται πως σε κάποιο στάδιο η εκπαίδευση ανδρών και γυναικών ε, αλλάζει την ε, περίοδο που ε, αποφασίζουν ε, τις, ε, τον κλάδο που θα ακολουθήσουν. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και κάτι ακόμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θέμα και σύμφωνα με τις εμπειρίες που άκουσα υπάρχει μάλλον το μία θα έλεγα <clears throat> έλλειψη βούληση των γυναικών για να ασχοληθούν με θέματα από τα μαθηματικά, ε, μηχανολογικά, γενικά. Ευχαριστώ. Mrs. Krebval, please. Ευχαριστώ. Από το Γυναικείο Λόμπι Και αυτά που μας είπατε δείχνουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ο κατακαιρματισμός, η διασπορά. Μιλάμε για ισότητα ανδρών γυναικών αλλά όχι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης και αυτό προκύπτει από τα στοιχεία. Λοιπόν, με τρόπο γενικότερο θα ήθελα να κάνω ε, μια διασύνδεση με την προηγούμενη παρουσίαση και το ζήτημα της οικονομικής ανεξαρτησίας διότι αυτά τα οποία λέτε για την εκπαίδευση δείχνουν τις τεράστιες επενδύσεις ε, που κάνουν οι, ε, τα κράτη-μέλη σε ό,τι φορά την εκπαίδευση των κοριτσιών και μετά όμως χάνονται όλα αυτά τα ταλέντα διότι δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες και διρωτώμε αν η εγγραφή στον προπολογισμό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να καταδεχθεί ναι, επενδύουμε, οι γυναίκες συμμετέχουν στην εκπαίδευση, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της επένδυσης που χάνεται διότι υπάρχουν τεράστιες ανισότητες σε επίπεδο μισθών, αμοιβών κλπ. Και έχουν γίνει μελέτες σχετικές για να καταδείξουμε το πώς επενδύσεις που γίνονται σε ζητήματα εκπαίδευσης κατάπεσης θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε οι γυναίκες να βγουν στην αγορά εργασίας και να οδηγήσει ως εκ τούτου στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Ευχαριστώ. Κυρία Μόλντερ, παρακαλώ να απαντήσει. Μικρόφωνο, παρακαλώ. Σχετικά με το πρόβλημα που θίξατε, ναι, όντως αναφέρθηκα Υπάρχουν ευθύνε ε, των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την διατύπωση των προγραμμάτων και την κατάρτιση, αλλά γνωρίζουμε επίσης ε, και η παρέμβαση του κυρίου το κατέδειξε πως εάν εμείς μένουμε ώστε η διάσταση του φύλου να συμπεριληφθεί, πολλά κράτη είναι ευαίσθητα σε αυτές τις ε, επιλογές. Και πιστεύω ότι όντως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Τώρα, αναφορικά με το ερώτημα, ειδικά με τις ε, επιλογές, έχετε εδώ στην Επιτροπή μια ομάδα που ασχολείται με το ζήτημα. Εγώ έχω ασχοληθεί με τα she figures του 2009 και φροντίζουμε να τα συνδυάσουμε με τις αποφάσεις του Ελσίνκη και να έχουμε ε, στοιχεία τεκμεριωμένα. Εμπεστούσει και αυτά τα στερεότυπα που αναφέρατε ότι υπάρχουν λιγότερες γυναίκες σε κάποιους κλάδους και όχι μόνο σε όλες τις ε, ερευνητικές ε, επιστήμες διότι υπάρχουν στον τομέα της βιολογίας περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες Γίνονται πάλι μελέτες που διεξάγονται σε επίπεδο επιτροπής ε, και παράλληλα χρηματοδοτούνται ε, κάποια ερευνητικά προγράμματα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε γιατί η πληροφορική, γιατί η μηχανολογία παραμένει ε, ένας τομέας σχεδόν αποκλειστικό ανδρικός αλλά βλέπουμε ότι σε άλλους κλάδους, π.χ. ιατρική, υπάρχουν πληθώρα γυναικών. Παραμένουν όμως αυτά τα σκληροπυρηνικά θα λέγαμε επαγγέλματα τα οποία συνεχίζουν να είναι όχυρα των ανδρών αλλά μελέτες διεξάγονται. Τώρα σε ό,τι φορά την ε, συμπλήρυψη της απασχόλησης ε, στην απασχόληση βλέπουμε ότι η ότι οι γυναίκες ε, σπουδάζουν, οι διαφορές μιστολογικές μισθολογικές, οι διαφορές της αμοιβές παραμένουν στάσιμες σε πολλά κράτη. Υπάρχει όμως και σύνδεσμο με αυτά που είχαμε πει στο παρελθόν ότι όταν θα σπουδάσουν οι γυναίκες αυτές οι διαφορές θα πάψουν να ισχύουν αλλά διαπιστώνουμε ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και στην αγορά εργασίας υπάρχει μια <clears throat> διτή θα λέγαμε ε, λειτουργία. Υπάρχουν γυναίκες που καταφέρουν να ακολουθήσουν στα διαδρομία και άλλες που δεν το κατορθώνουν. Ευχαριστώ κυρία Μιούλντερ για την παρουσίαση. Περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μισθές διατάξεως. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λιμπεράκη που θα μας παρουσιάσει ανάλυση για την υγεία, την ευμερία για το περιβάλλον όπως και οι υπόλοιποι αγορητές έχετε 15 λεπτά για την παρουσίαση ξέρω πως ε, είναι δύσκολο να περιοριστείτε διότι έχετε δουλέψει πολύ καιρό αλλά παρακαλώ αν μπορείτε να παραμείνετε εντό 15 λεπτού, σα ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Όταν εξετάζουμε το ζήτημα της ιδείας, ε, του περιβάλλοντος και της ευημερίας, το πρώτο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό μας είναι ποια είναι η σημασία αυτού του θέματος από πλευράς ε, ισότητας ε, των φίλων. Η προσέγγιση λοιπόν που ακολουθήσαμε δείχνει ότι ε, αυτή η τομή είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα της ζωής των γυναικών αλλά μπορούν να αποτελέσουν και την πηγή ανισοτήτων μεταξύ των φίλων τόσο άμεσα όσο και, άμεσον όσο και έμεσον. Γνωρίζουμε, και αυτό τονίστηκε σε προηγούμενες ομιλίες, ότι στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος, της ευημερία ε, και της ευεξίας, ε, ε όλα αυτά είναι θέματα που αρμπίπτουν αρμοδιότητες των κρατών μελών. Φυσικά υπάρχει η επικουρικότητα που ισχύει και ε, όμως αυτά τα οποία συμβαίνουν αποφασίζονται σε χαμηλότερο επίπεδο. Με όλα τα αυτά όμως είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά δηλαδή να έχει μια έμμεση επιρροή με ε, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πολύ ευρύτερο από ό,τι μας λένε τα στοιχεία τα καθεαυτά. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, σχετικά μικρά κονδύλια αλλά να έχουμε ευρύτερες ε, επιπτώσεις, ευρύτερο αντίκτυπο στους τομείς αυτούς. Μια άλλη δυσκολία όταν ε, μιλάμε για την ευημερία των περιβάλλων, την υγεία σε σχέση με την ισότητα των φύλων, ότι πολλοί από τους στόχους έχουν την νόημα του δημόσιου χαρακτήρα. Και πολλά αυτά που ε, οι οικονομολόγοι αναφέρουν ως additionalities, προσθετικότητες, ε, λειτουργούν Λοιπόν, όσο πιο μακροπρόθεσμος είναι ο ορίζοντας ο στόχος, τόσο λιγότερο ακριβής μπορεί να είναι η αξιολόγηση του αντικτύπου. Το βασικό στοιχείο της παρουσίασής μου θα αφορά αυτούς τους τρεις στόχους. Πολλοί στόχοι τίθενται αλλά με τρόπο ιδιαίτερα ευρύ, αφηρημένο θα λέγαμε. Και η άλλη πλευρά είναι πως ε, ίσως ε, να ε, φτάσει το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να αναλάβουμε κάποια δράση. Τώρα, στο θέμα της υγείας και των φίλου η καλή ή η κακή υγεία μπορεί να ε, έχει άμεση επίπτωση στην ε, ισότητα των φύλων. Τώρα, ποιοι εργάζονται στον τομέα της υγείας, την πλευρά της προσφοράς. Αν κάνουμε την κατανομή μεταξύ ανδρών γυναικών στον κλάδο, βλέπουμε ότι οδηγούμε σε μια πόλωση. Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στον τομέα της ε, νοσηλευτικής ε, ενώ οι άντρες ε, έχουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε ιατρικά επαγγέλματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην, ε, ε, στην περίθαλψη και στις ιατρικές υπηρεσίες, ε, φυσικά έχουμε και το οικονομικό ζήτημα που διαδραματίζει ρόλο, αλλά έχουμε και κάποιες ειδικές ομάδες όπως μετανάστες ε, άτομα αποκλεισμένα από την κοινωνία, γυναίκες κλπ. κλπ. Σε ορισμένες περιστάσεις, περιπτώσεις, αυτές οι κατηγορίες συμπίπτουν. Τώρα, αφορικά με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, τι κάνουμε για να είναι το δυνατόν καλύτερη η υγεία των πολιτών, βλέπουμε ότι η χορήγηση πόρων σε ειδικέ ε, συνθήκες δεν είναι ίση και ισότιμη. Δεν έχουμε τις ίδιες ε, συνθήκες. Αυτό σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την ε, δυνατότητα επιρροής ε, ενός ε, υγιού τρόπου διαβίωσης, health lifestyle. Τώρα, ο στόχος του εγγράφου στρατηγικής ε, να φέρει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ανισότητες των φύλων τουλάχιστον αυτές που είναι προβλέψιμες. Και αυτό εξαρτάται φυσικά από το πόσα κονδύλια θα διαθέσουμε σε συγκεκριμένες ασθένειες κλπ. Μερονώ ότι άνδρες και οι γυναίκες γυράσκουν για να κάνουμε όλοι μεγαλώνουμε και όλοι γνωρίζουμε πως ε, οι γυναίκες ε, είναι μακροβιότερες ε, των ανδρών. Αυτό δεν είναι πάντα θετικό. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα όπου στο πάνω κομμάτι βλέπετε την κατανομή ανδρών με μπλε, γυναίκες με κόκκινο σε ευρωπαϊκά κράτη Ε, προσώπων ηλικία άνω των 50 που πάσχουν από δύο ή παραπάνω χρόνιες ασθένειες. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ είναι πως σε κάθε κράτος ε, που αναφέρεται στο παράδειγμα οι γυναίκες τείνουν να πάσχουν περισσότερο ως ποσοστό του πληθυσμού σε σύγκριση με τους άντρες από δύο ή περισσότερες χρόνιες ασθένειες. Το κάτω γράφημα δείχνει ε, πρόσωπα με κλινικά ουσιαστικές ε, ε, κατάθλιψη και εδώ βλέπουμε ότι η διαφορά είναι πιο σαφής. Μόνο ότι οι γυναίκες ε, ζουν περισσότερα χρόνια, αλλά ε, υποφέρουν από περισσότερες ε, χρόνιες παθήσεις και δι κατάθλιψη. Και αυτό ε, ισχύει για όλα τα κράτη. Τώρα, σχετικά με την ευημερία, ακόμα και στις κοινωνίες με οικονομία την αγορά, όπου υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε πόρους και σε χρήμα, Ε, υπάρχουν ε, λόγοι όπως ε, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης και σε σε μια πιο περίπλοκη και διαφρομένη κοινωνία. Και εδώ ε, οι γυναίκες εμπλέκονται διότι ασχολούνται, μελοφέρουν αυτό το διτό άχθος, δηλαδή ασχολούνται με την οικογένεια, ε, εργάζονται, φροντίζουν τα παιδιά κλπ. Και θεωρούμε λοιπόν ότι η προστασία του καταναλωτή μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις ε, στην ε, ευημερία των γυναικών. Τώρα, ε, ευημερία είναι ένα θέμα πιο περίπλοκο και εδώ θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τώρα, ένα στοιχείο για την ευτυχία που έχουμε για την ευτυχία των γυναικών ε, παρατηρούμε ότι ε, τα τελευταία 30 χρόνια η ευτυχία ε, στις γυναίκες έχει μειωθεί και επίσης υπάρχουν, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα φύλλα σχετικά με το χρήματα τα οποία διαθέτουν και την ευτυχία. για τα, με το ίδιο ποσό οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες. Αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα. Υπάρχουν διαφέρουσες όμως ερμηνείες, αλλά προφανώς πολλά μπορούν, απομένουν να γίνουν σε αυτό το τομέα και αυτό το είδος προσέγγιση αφορά άμεσα την ε, ισότητα των φύλων. Τώρα, επανερχόμενοι στο περιβάλλον, ε, η πλευρά της προσφοράς, της προμήθειας. Το περιβάλλον είναι στο τομέας που θα προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας στο μέλλον. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τις διαφορές ανάμεσα στα φύλλα αλλά και επειδή είναι ένας τομέας ε, εντάσσεως κεφαλαίου είναι προφανές ότι οι γυναίκες θα δυσκολευτούν να αναλάβουν παρόμοιες δραστηριότητε σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό συνδέεται και με το θέμα των δημοσίων μεταφορών, τη βελτίωση αυτών, κάτι το οποίο έμεσα μπορεί να επηρεάσει τις γυναίκες ως τους ε, βασικούς χρήστες. Και υπάρχουν όμως και ζητήματα ασφάλειας, πρόσβαση στις αστικές περιοχές Όλα αυτά είναι τομείς σε έναν ευρύτερο πίνακα που μπορούν άμεσα ή έμεσα να επηρεάσουν τις σχέσεις των φίλων, αλλά δύσκολα μπορούμε να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. Λοιπόν, από τη στρατηγική στην εφαρμογή τα τρία βήματα. Πρώτα, ανάλυση των στόχων, τι πρέπει να γίνει. Δεύτερον, τι μας λένε τα έγγραφα της Ένωσης και περνώντας ε, στον προπολογισμό, το κοινωνικό ταμείο και άλλα. Θα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα προβλήματα ε, ισότητας του φύλου θα πρέπει να ε, δούμε τι θα συμβεί μέχρι το 2020 αν ε, συγγνώμη κάποιο πρόβλημα έχω με την οθόνη μου βλέπετε λοιπόν τον προπολογισμό για τον υγεία των περιβάλλον ε, και Εάν πάτε στην κάτω γραμμή θα δείτε τις αλλαγές ε, σε σχέση με τους προηγούμενους προπολογισμούς ε, και αυτέ ε, είναι πολύ σημαντικές, πολύ περισσότερους πόρους σε όλους σχεδόν τους κλάδους εκτός από την γεωργική πολιτική και ουσιαστική αύξηση των πόρων στον τομέα της έρευνας. Και προς το παρόν όμως δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ε, στην ισότητα των φύλων. Και τώρα να περάσω τα συμπεράσματα λέγοντα ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να επαγρυπνούμε. Οι πρώτοι στόχοι που αφορούν ε, την υγεία, περιβάλλον κλπ ε, απαιτούν νέες ε, δεξιότητες. Τώρα το αυτή η τύφλωση θα λέγαμε των φίλου μπορεί να, διακινδυνεύσει, την ισότητα του φίλου και τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας κλπ. Και οι πράσινες ε, θέσεις εργασίας ε, πρέπει να είναι ουδέτερες ε, σε ό,τι αφορά τα δύο φύλλα. Ο τομέα της ενέργειας και της υγείας θα είναι από τους κύριους κλάδους Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε, να στοχεύσουμε μάλλον στην ισότητα των φίλων σε αυτές τις ε, δύο δράσεις. Και αν διορθωτικές ε, δράσεις δεν αναλυφθούν έγκαιρα, δίχως ε, να ελέγξουμε και να εποπτεύσουμε τους ε, τομείς αυτούς αποτελεσματικά, τότε ενδέχεται να καταλήξουμε στο να επιταθούν οι ε, διαφορές ανάμεσα στα φύλλα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και θα ήθελα να ε, μου πείτε αν υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. No questions, no... Oh, sorry. Mrs. Glass, please. Κύριε Κλάς. Με συγχωρείτε, έπρεπε να πάω κατά σε μια άλλη συνεδρίαση. Αλλά αυτά που άκουσα τώρα στο τέλος ε, με κάνουν πιστεύω ότι επανερχόμαι σε αυτό που είχα πει εγώ αρχικά. Δηλαδή πώς μπορούμε τώρα στον τομέα του περιβάλλοντος, στο κοινωνικό τομέα, να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τις γυναίκες και να πούμε τώρα θα έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για τις γυναίκες. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος και όσον αφορά θέματα κοινωνικά ή και προπολογιστικά αν θέλετε. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μέλος και ξέρω ότι οι γυναίκες στον τομέα της ενέργειας είναι πάρα πολύ ευαίσθητες, γιατί το 40% της ενέργειάς μας έτσι και χρησιμοποιείται στα νοικοκυριά. Και ψάχνω τώρα να βρω πώς θα μπορούσα εδώ συγκεκριμένα να βρω κάτι για τις γυναίκες, ούτως ώστε να μπορέσουν πραγματικά να έχουν ε, μια άμεση πρόσβαση. Περίμενα η δική σας παρουσίαση να μας ε, ε, βοηθήσει εκεί. Τι μπορούμε να κάνουμε, να ετοιμάσει το Κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα για τις γυναίκες ούτως να μπορούσαν να δράσουν ιδιαίτερα επειδή είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες και επειδή έχουν και τις γνώσεις και επειδή μπορούν να ενημερώσουν από εκεί και πέρα. Ίσως θυμάστε κύριε Πρόεδρε ότι στο, στα πλαίσια της έκθεσης για το κλίμα είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τις γυναίκες στον τομέα του κλίματος, του περιβάλλοντος να δράσουν, αλλά δεν ξέρω πού μπορώ να βασιστώ. Μήπως μπορείτε κάτι να μου πείτε πάνω σε αυτό. Να με βοηθήσετε. Πρώτος, θα δώσω το λόγο στην κύριε Λιμπεράκη. Okay. What I tried to show... Αυτό που προσπάθησα να σας δείξω στην παρουσίασή μου ήταν ότι σε αυτούς τους τομείς, παρόλο που όλοι κατανοούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στην ε, ποιότητα της καθημερινής ζωής. Είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσει κανείς με ακρίβεια την ε, ε, διάσταση φύλου. Αυτό δεν ισχύει ίσως για την υγεία και γι' αυτό σας έδειξα ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ασθένειες και κακή υγεία και όσον αφορά την φυσική τους υγεία και όσον αφορά προβλήματα πνευματικής υγείας. Λοιπόν, αυτή είναι μια δυνατότητα για να ορίσουμε τα διάφορα προβλήματα και η άλλη μεριά είναι να δούμε ποιος εργάζεται σε αυτούς τους τομείς. Και εδώ υπάρχει μια δυνατότητα απάντησης ε, για να δώσουμε μια σαφή ε, διάσταση του φίλου. Ποιο εργάζεται δηλαδή σε αυτούς τους νέους τομείς, στα νέα σχέδια με τις νέες αυτές επενδύσει όσον αφορά την υγεία, την ευημερία και το περιβάλλον. Ομολογώ βέβαια ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, είμαι κάπως σκεπτικιστής και πρέπει να σας το πω ξεκάθαρα. Όταν συνεχώς λέμε ότι οι γυναίκες συσχετίζονται με την κατανάλωση ή με τη λήψη αποφάσεων στα νοικοκυριά, όχι επειδή το αρνούμε ότι πραγματικά οι γυναίκες συνοικίες που καταναλώνουν κυρίως ε, όπως παράγουν σε μεγάλα τμήματα του κόσμου αλλά αυτό ε, είναι ένα στερεότυπο κατά κάποιον τρόπο Θα πρέπει βέβαια να δώσουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες όταν αποφασίζουν για οτιδήποτε αποφασίζουν να είναι ενήμερες οι αποφάσεις τους και θα πρέπει να ξέρουν ποιες είναι οι επιπτώσεις των αποφάσεων που παίρνουν. Αλλά είναι σαφές για με ότι δεν είναι οι γυναίκες εκείνες οι μόνες που αποφασίζουν για την κατανάλωση. Παρόλο λοιπόν που βλέπω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έμεση ή άμεση επίπτωση στις γυναίκες, παρόλα αυτά ελπίζω στο μέλλον, δεν ξέρω πόσο εγγύς θα είναι το μέλλον αυτόν ή απόμακρο, θα εξαφανιστούν αυτοί οι συσχετισμοί ορισμένης, ομα... ορισμένης ομάδας ατόμων με κάποια στερεότυπα. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποιος προσλαμβάνεται. Αυτό είναι εύκολο να δει. Στην έρευνα, στην κοινοτομία, στο περιβάλλον κλπ. Και δεύτερον να δούμε ποιος ωφελείται από την κατάσταση αυτή. Και είναι σαφές ότι αν κανένας κάνει έρευνα για, την, ε, για το καρκίνο του μαστού, ξέρει ποιος ωφελείται. Και αν κάνει έρευνα σε έναν άλλο τομέα και είναι επιτυχής η έρευνα αυτή, πάλι ξέρει ποιον στον ωφελεί. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν, πολλά που δεν ξέρουμε πολλά που πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Ξέρουμε όμως αρκετά για να μπορέσουμε να πάρουμε πιο αποφασιστικές δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, έχω και εγώ μια ερώτηση. Θα σας την υποβάλω στα σουηδικά γιατί είναι πιο εύκολο για μένα. Είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανένα κάποια θέση, κάποια ισχύ στην αγορά απασχόλησης. Είναι πραγματικά σημαντικό να δει κανένας πώς παίρνει κάποιος και με ποιες δομές τις αποφάσεις. Στον τομέα των μεταφορών, Φερρυπίν, μπορούν άντρες και γυναίκες να κινούνται εκεί και ελπίζω να είναι ισότιμα αυτή η κίνηση στο μέλλον. Σήμερα όμως η κίνηση δεν είναι η ίδια αν είναι κανένας άντρας ή γυναίκα, διαφέρει ο τρόπος μετακίνησης. Παραδείγματος χάρη, οι γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα μαζικών μεταφορών, οι άντρες περισσότερο με γιοταχή. Όταν λοιπόν αποφασίζονται υποδομές, χρειάζεται κάποιος λέγεται όμως περισσότερους δρόμους και όχι ενίσχυση των ε, ε, δημοσίων μέσων μεταφοράς, ε, μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πού λαμβάνονται και πώς λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις. Αυτό έχει σημασία ήδη σήμερα. Κατά πόσο θα επενδύσει κανένα ε, μέσα μαζικής μεταφοράς ή θα επενδύσει αυτοκινητόδρομους. Αυτό στο μέλλον θα είναι το ίδιο ή όχι. Αλλά η κυρία Αντάρ έχει το λόγο. Ναι. Αυτό που ακούμε με έκανε να σκεφτώ ποιες είναι οι οικονομικές αποφάσεις που παίρνουν οι γυναίκες σε όλους τους τομείς. Η οχι αλλα η κυρια δεν εχει το λογο ναι αυτο που ακουμε με εκανε να σκεφτω ποιε ειναι οι οικονομικέ αποφάσει που παιρνουν οι γυναικες σε ολους τους τομεί. υγεια περιβαλλον την, ε, διορδομία του, στη δουλειά του, αυτή τη γενική εικόνα. Και το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα είναι το εξή. Ξέρετε όλοι ότι η Ιδανική Προεδρία τονίζει το ρόλο των γυναικών στι κλιματικέ αλλαγέ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τη εργασία που θα γίνει στου επόμενου έξι μήνες που ίσως τελικά οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του ρόλου των γυναικών στο περιβάλλον όχι μόνο στις κλιματικές αλλαγές, αλλά και σε άλλους τομείς του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η κυρία Λιμπεράκη για να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές σας και τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν, ε, κύριε Πρόεδρε, γιατί πραγματικά θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Ότι εκείνος που παίρνει την απόφαση έχει επίδραση πάνω στην παρφή της απόφασης. Η διαδικασία λοιπόν ύψης αποφάσεων έχει να παίξει ένα πολύ ρημανικό ρόλο. Και επίσης το γεγονός ότι οι αποφάσεις επέρνοντο όπως επέρνοντο έχει επιδράσει στα όσα έχουν ενωθεί μέχρι στιγμής. Αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και προτεραιότητες. Θα πρέπει λοιπόν να ε, στοχεύσουμε και στις διαδικασίες λήψης αποφασής και στις προτεραιότητες. Όσον αφορά το ρόλο των γυναικών στις κλιματικές αλλαγές, υπάρχει νομίζω έντονη συζήτηση για το θέμα αυτό. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής ομολογώ είναι κάπως πτωχά. Αλλά βέβαια θα πρέπει να παραμένει κανείς ενδεμένος με αυτό που συζητούνται. Γιατί ελπίζουμε ότι αυτά θα οδηγήσουν σε πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από αυτά που σήμερα θεωρούνται αυτονόητα πριν από λίγο καιρό θεωρούνται τελείως ε, ουτοπικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λιμπεράκη. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Και θα ήθελα εδώ να καλωσορίσω την κυρία Ράβερη που θα μας κάνει μια παρουσίαση σχετικά με τα βασικά δικαιώματα. Έχετε και εσείς 15 λεπτά για να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα και την ανάλυση σας. Okay, thank you. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσίαση μου αφορά το ρόλο της ε, Χάρτας Βασικών Δικαιωμάτων στην ισότητα των φύλων καταρχήν και κατά δεύτερον πώς ε, το πολιετές ε, δημοσιονομικό ταμείο συμβάλλουν στην λήψη υπόψη των, της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και στο mainstreaming για τα βασικά δικαιώματα. Όπως γνωρίζετε, η Χάρτα των Βασικών Δικαιωμάτων διακρίθηκε το 2000 και τέθησε νομικά δεσμευτική μορφή το 2009 μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει εκεί ένα κεφάλαιο ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους ε, τομείς συμπληρωμένως ε, εργασίας, απασχόληση και μισθού και επίσης το δικαίωμα της μη διάκρισης, αρνητικής διάκρισης. Άμα δούμε τι μας δίνει η χάρτα αυτή σαν ε, βάση για την πρόθεση της ισότητας των φύλων, μπορούμε να έχουμε κατά νου κάποια πολύ σημαντικά σημεία. Παραδείγματο χάρη επαναβεβαιώνει την δέσμη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Και αν εξετάσει κανένας αυτά τα πολιτή προγράμματα και την χρηματοδότηση για την ισότητα, ε, πρέπει να έχουμε κατά νου την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μεγάλο τμήμα τη προστιθέμενης αξίας είναι ακριβώς η ισότητα των φύλων που προωθήθηκε και σε χώρες που δεν είχαν τέτοιες προτεραιότητες στο παρελθόν. Είναι λοιπόν πολύ ε, σημαντικός ο ρόλος της χάρτας για την προώθηση των δικαιωμάτων αυτών. Τα δικαίωμα για μη διακριτικές ε, ε, μεταχείρισεις όπου ισχύει και για τα δικαιώματα ατόμων από τρίτες χώρες βλέπουμε ότι αυτό είναι ε, όχι μόνο οι γυναίκες έναντι των ανδρών σαν ομάδες διαφορετικές μεταχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε περισσότερα πραγματικά το γεγονός ότι η, η φτώχεια είναι όσο πάει και γίνεται και πιο γυναικεία ή και η μετανάστευση. Επίσης η χάρτα αυτή ο... αναγνωρίζει ότι υπάρχει εμπόριο ε, ανθρώπων σε μεγάλο μεγάλο βαθμό Πράγμα που αποτελεί βέβαια μια παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τέλος δίνει τα δικαιώματα των πολιτών και το δικαίωμα της ισότητας ενώπιον της δικαιοσύνης και δίνει τη δυνατότητα έτσι να μπορούν όλοι να προωθήσουν την ισότητα των φίλων. Εγώ τώρα θα θέλω να περάσω αυτό που δεν κάνει η κάρτα αυτή, γιατί η κάρτα αναφέρει τις λεγόμενες ανητικές ελευθερίες. Δηλαδή ζητά ε, να μην υπάρχουν κάποια εμπόδια και περιορισμοί στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην εργασία, στην απασχόληση κλπ. των γυναικών. Αλλά θα πρέπει αυτές οι αρνητικές ελευθερίες να γίνουν θετικές ελευθερίες, δηλαδή να δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχουν προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δυνατότητα αυτή της άσκησης των δικαιωμάτων τους και θετικέ ελευθερίες βλέπει ότι υπάρχουν τρεις, α, τρία πράγματα απαραίτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχήν ευρωπαϊκή και χρηματοδότηση για να συνεχίσουμε να προωθούμε και να υποστηρίζουμε την ισότητα των φύλων σαν μια κοινή αξία όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης χρειαζόμαστε πιο σφαιρική προσέγγιση στην πολιτική που εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του λεγόμενου ε, mainstreaming. Δηλαδή για να μπορούν οι γυναίκες ε, να ε, πάνε να εργαστούν χρειάζεται κάποιος να φροντίσει τα παιδιά τους. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσει κανένας ότι αν περικόψει κανένας την φροντίδα αυτή των παιδιών όπως είπε και η κυρία Μπέτιο, υποσκάπτει το δικαίωμα τη γυναίκας να πάει να εργαστεί. Επίσης χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, ούτω ώστε να ξεπεραστούν συγκεκριμένα εμπόδια και περιορισμοί και να δώσει τη δυνατότητα άσκηση των δικαιωμάτων και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, τα θέματα αυτά τη μη ισότητα των φύλων να είναι ορατά. Και ένα πρόβλημα είναι ότι αυτό το θέμα του φύλου δεν είναι πια τόσο ορατό. Μέσω της ανάλυσης αυτής λοιπόν είδαμε κάποιους βασικούς στόχους ε, που βασίζονται στα βασικά δικαιώματα, στη χάρτα των βασικών δικαιωμάτων. Καταπολέμηση της βίας, του εμπορίου των ανθρώπων, ισότητα ανθρώπων και ε, ανδρών και γυναικών όσον αφορά την ίση αμοιβή, η ισορροπία όσον αφορά την διαδικασία λήψης απόφασης, ε, καταπολέμηση της φτώχειας και της μετανάστευση και μέτρα που δίνουν τη δυνατότητα των όρων για την πλήρη άσκηση των βασικών δικαιωμάτων δημοκρατικής συμμετοχής, δικαιοσύνη όταν ενώπιον της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Στρεφόμενοι τώρα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, όπως αναφέρθηκαν, κοιτάξει κανένας τα έγγραφα, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό που δεν αναφέρεται καθόλου το mainstreaming του φίλου και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια για την πρόθεση της ισότητας. Θα έπρεπε όμως αυτό να είναι ένας οριζόντιος στόχος όλων των προγραμμάτων και γι' αυτό η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον γενικό κονοσμό είναι ένα πρόβλημα. Για να αποφύγουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αναλύσουμε τα συγκεκριμένα προγράμματα που είναι ουσιαστικά για την Χάρτα των Βασικών Δικαιωμάτων και εκεί βλέπουμε τρία, δηλαδή το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την, ε, τα πολιτικά δικαιώματα. που υπάρχουν τα προγράμματα Δάφνη 3, βασικά δικαιώματα και ε, πρόγραμμα για ισότητα των Φίλων και κατά των διακρίσεων και υπέρ της διαφορετός. Επίσης ε, υπάρχει εδώ το Ταμείο για την μετανάστευση και το άσυλο. Αν δει κανένα ε, τα έγγραφα που υπάρχουν και το προβολισμό που υπάρχει από κάποια φύλου, θα πρέπει να δούμε το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ε, <clears throat> δικότητα. Τώρα ελήφθη μια απόφαση να ενσωματωθούν αυτά τα τρία προγράμματα που σας προανέφερα αλλά το τμήμα της ισότητας του προγράμματος Progress που αφορούσε ακριβώς στόχους ε, για την ισότητα. Έχουμε το Δάφνη 3 που είναι ε, κατά της βίας και των παιδιών και ένα άλλο πρόγραμμα που έχει συγκεκριμένο στόχο την ισότητα των φύλων. Τώρα βλέπουμε να μην υπάρχει ενημέρωση όσον αφορά τον προπολογισμό του νέου αυτού προγράμματος που ενσωματώνει τα τρία προγράμματα που σας προανέφερα. Δεν υπάρχουν υποδιαιρέσεις, δεν έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποσά που θα δαπανηθούν μέσα στα πλαίσια των διαφόρων αυτών συνοστισών. Για το πρόγραμμα 2007-2013 το Δάφνη υπήρχε μια καλή απόδοση. Το πρόγραμμα των βασικών δικαιωμάτων βλέπουμε ότι δεν έχει καμία αναφορά στο φύλλο. Η μόνη εξαίρεση είναι η υπηρεσία για τα βασικά δικαιώματα όπου στην ετήσια της έκθεση αναφέρεται πολύ καλά και το θέμα του φύλου και όπου υπάρχει ένα ε, ξεχωριστό κεφάλαιο για το φύλο ιδίως ε, το κεφάλαιο που αφορά τους Ρωμά που τονίζει ιδιαίτερα τις γυναίκες είναι λοιπόν ε, μια έπληξη που το σφαιρικό πρόγραμμα σχεδόν δεν αναφέρεται καθόλου στο φύλλο, ενώ ο οργανισμός, ε, ο αρμόδιος, το κάνει. Ε, όμως το αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενσωματώνοντας τα τρία αυτά προγράμματα, το ένα από τα οποία δεν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα φύλου, έχουμε τον κίνδυνο το φύλλο να είναι λιγότερο ορατό και να δαπανούνται και λιγότερα χρήματα γι' αυτό γιατί ένα από τα κίνητρα για την ολοκλήρωση ήταν ακριβώς η δυνατότητα μεταφοράς ποσών μεταξύ των τριών αυτών προγραμμάτων. Και στο τέλος ομιλίου θα το ξανασχολιάσω αυτό. Είναι επίσης ε, ορατό ότι το... ο προπολογισμός μειώθηκε στο 95,6% του προηγούμενου προπολογισμού. Το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί προωθεί την κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή όλων. Έχει μειωθεί και εκεί ο προπολισμός, αλλά οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την προώθηση της ε, ατζέντα για την ισότητα και για τα βασικά δικαιώματα. Δεν αναφέρεται ρητά το φύλλο, Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σημαντικά στοιχεία στα οριζόνια, στην οριζόνια παρουσίαση του προγράμματος του 2007-2013 που όχι μόνο καλούν για ισότητα των φύλων αλλά ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. Γιατί βέβαια αν γυναίκες δεν είναι σε ένα πρόγραμμα δεν θα εμπλακούν. Δεν έχω δει ακόμα τα έγγραφα για το 2014-2020 για το πρόγραμμα αυτό. Ελπίζω όμως ότι θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή. Δυστυχώς όμως δεν συμπεριλαμβάνει το φύλλο και συγκεκριμένους στόχους στα θεματικά κεφάλαια για τα επόμενα έτη. Είναι καλό λοιπόν αλλά δεν είναι πιστικό και επίσης το νέο ταμείο για την ε, ε, μετανάστευση και το άσυλο δεν βρήκαμε καμία αναφορά σε ισότητα των φύλων. Θα ήθελα λίγο να περάσω σε κάποιες συστάσεις και συμπεράσματα. Είπαμε ότι το ε, πρόγραμμα δημοσιονομικού πλαισίου δεν αναφέρει καθόλου την ισότητα ή το mainstreaming. Επίσης όσον αφορά τα προγράμματα Δάφνη ή εκείνο που αφορά τα βασικά δικαιώματα επίσης μειώνουν την ορατότητα του, της του φύλου. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι. Καταρχήν ότι θέματα της ισότητας των φύλων θα εξαφανιστούν μέσα σε γενικά θέματα κατά των αναλυτικών διακρίσεων, αλλά το θέμα του φύλου δεν θα είναι πια τόσο ορατό και απουσία συγκεκριμένων προπολογισμών για το φύλλο βασιζόμαστε στο gender trimming, στο mainstreaming δηλαδή του, της διάστασης του φύλου. Πολλοί το ξεχνάνε όμως αυτό. Υπάρχει μια γενική δέσμευση για κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι όλοι το ξεχνάνε αυτή τη στιγμή. Και ούτε ακολουθείται, ούτε επαρκεί από μόνο του αυτό. Και επίσης υπάρχει, εκτός από τη μείωση στο συνολικό προπολογισμό, υπάρχει ο κίνδυνος τα χρήματα να φύγουν από θέματα που αφορούν μόνο τα φύλλα, εάν η ισότητα των φύλων δεν είναι μία από τις πολιτικές ε, προτεραιότητες των επόμενων ετών. Για να μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα που έχουμε ήδη αναφέρει σήμερα δηλαδή να υπάρχουν άμεση και βατή στόχοι για την ισότητα με τους σωστούς και προβλέπιμους προπολογισμούς, προς υιοθέτηση διτής προσέγγισης για το mainstreaming, συμπληρώνονται με συγκεκριμένες δράσεις οποιασδήποτε ανισότητες υπάρχουν μεταξύ άνθρωπων και γυναικών, εποπτεία και αξιολόγηση των επιπτώσεων των ε, δημοσιονομικών, της δημοσιονομικής εφαρμογής ε, για την ισότητα των φύλων και συμπεριλαμβανομένων και των στατιστικών στοιχείων που θα χωρίζονται ανά φύλλο. Χωρίς να πρέπει κάποιος να αποφασίζει αν κάθε φορά αυτό είναι σημαντικό ή όχι. Και ε, ο έλεγχος και η υποπτία της πραγματικής χορήγησης ε, του προπολογισμού για τα δικαιώματα και την ε, ιδιότητα του πολίτη για την ισότητα εφόσον δεν υπάρχουν νέοι συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν ξέρω. Μήπως τώρα πρέ... πρόκειται να μειωθεί το ποσοστό που δίνεται την ζητότητα των φίλων. Επίσης εξετάσουμε πώς θα, εξετάσουμε, πώς θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς μέσα στα πλαίσια μιας ε, πολιτικής λιτότητας. Αναφέρθη ότι οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα ε, ρίχνουν την ισότητα των δύο φύλων στα περιθώρια της ε, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να αναγνωρίζετε ότι αυτό δεν είναι κάτι που είναι πολυτέλεια αλλά το θέμα της ισότητας είναι βασικό θέμα και η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόθεση της ισότητας των ε, ε, φίλων είναι τόσο σημαντική που θα πρέπει να δούμε πώς προωθούνται οι δυνατότητες των γυναικών για την άσκηση των βασικών τους ε, δικαιωμάτων. Παραδείγματο χάρη είπα προηγουμένως, αν κάποιο ε, θέλει να εργαστεί, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα φροντίδα του παιδιού του. Αν περικοπούν αυτά τα προγράμματα της φροντίδας παιδιών, μειώνεται το βασικό δικαίωμα της γυναίκας να εργαστεί. Επίσης το θέμα των ευελίκτων προϋπολογισμών ίσως οδηγεί στο κανένας να μην εξετάζει ποιες είναι οι επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής κρίσης στις γυναίκες. Πολλά ελέγξαν για την άμεση επίπτωση της οικονομικής κρίσης του 2008 στην απασχόληση των ανδρών γιατί δεν υπάρχει πια τόση πολλή εργασία στον ε, τομέα των οικοδομών ή της ε, ε, παραγωγής κλπ. Εάν δεν κάνουμε κάτι παρόμοιο για να ελέγξουμε τις επιπτώσεις των περικοπών στο δημοσίου τομέα που θα έχουμε τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος η ισότητα των γυναικών να παραμείνει σε χαμηλό επίπεδο προτεραιότητας της πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε σαφές ότι χρειάζεται να μειωθούν οι επιπτώσεις της ε, κοινωνικής ε, ανισότητας και τέλος έχοντας ακούσει μερικούς που ζήτησαν να υποβάλουν ερωτήσεις, ε, θέλουμε, λέω, να προωθήσουμε την κοινωνία των πολιτών, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προωθηθεί η ισότητα των ε, φίλων και να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να συμμετάσχουν στην πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 που αν οι γυναίκες δεν συμμετάσχουν δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προωθηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρούμπερ, και τώρα ακούμε ερωτήσεις, σχόλια. Yes, please go ahead. Yeah, hi. Uh, my name is... Εκπροσωπώ εδώ το Ευρωπαϊκό Λόμπι των Γυναικών και ονομάζομαι Anne Wintermeers. Θα ήθελα να σε ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και την ε, επισήμανση των προβλημάτων που έχουμε δει και εμείς από πλευράς μας στο Ευρωπαϊκό Λόμπι των Γυναικών. Κάποια προβλήματα ωστόσο. Μιλήσατε για αποκλήσει ω προ τα συνολικά ποσά τα οποία διατίθενται για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων και είπατε ότι μπορεί οι ανισότητες να είναι υψηλότερες 30% κτλ. Επίσης μας ανησυχεί ιδιαίτερα το τι επιφυλάσσεται μάλλον για το πρόγραμμα Δάφνη. Η ισότητα ε, όχι μόνο δεν υπάρχει στους στόχους της Επιτροπής ως γενική πολιτική, αλλά ούτε και ιδιαίτερη διάσταση για τις γυναίκες δεν προβλέπεται. Και έτσι θέλουμε τουλάχιστον οι δραστηριότητε του προγράμματος Δάφνη να συνεχίσουν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Τελευταία μου παρατήρηση. Είναι άκρο ε, σημαντικό τις συζητήσει που γίνονται, θα γίνουν τώρα την άνοιξη, να τι αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσει την πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται για μια πρόταση μόνο, μπορεί να αλλάξουν αρκετά πράγματα, υπάρχει περιθώριο για τροποποίηση, για βελτίωση πολλών πραγμάτων. Πολλή δουλειά μένει να γίνει λοιπόν. Και έτσι παρακαλώ την κυρία Ζούμπερ τώρα. λόγο. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εισήγησή σας. Ιδιαίτερος. Σε σχέση με ένα ζήτημα που ετέθη προς το τέλος. Την περιγραφή δηλαδή του σωστού πλαισίου για συγκεκριμένη αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με το φύλλο μέσα στα δεδομένα της ε, κρίσης. Και τώρα ερωτήματα που έχουμε διατυπώσει και στο παρελθόν πρέπει να τα αναδιατυπώσουμε. Γιατί η κρίση και η πολιτική της λιτότητας επηρεάζει τα πάντα πλέον. Έτσι, θα ήταν πιστεύω απαραίτητο ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την ειδική, την ειδική χρηματοδότηση έτσι ώστε αυτές οι ανισότητες να αντιμετωπιστούν ακόμη πιο στοχευμένα. Διότι τουλάχιστον από τη δική μου τη σκοπιά η πολιτική λιτότητας οδηγεί σε περικοπές, οδηγεί σε ε, είτε διακινδύνευση είτε εγκατάλειψη μια σειρά από κοινωνικά και ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ε, παραβλέψουμε τις ε, συνέπειες, των αντίκτυπων που μπορεί να έχουν αυτά τα μέτρα λιτότητας. Εγώ παίρνω σαν παράδειγμα βέβαια την πατρίδα μου, είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να απολύσει ο εργοδότης τους εργαζομένους του. Και βέβαια αυτό έχει συνέπειες σε κάθε άλλο δικαίωμα του εργαζομένου, εφόσον μπορεί να τον απολύσει κανείς τόσο εύκολα. Και πάντα πληττόμενες περισσότερο είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων. Και μπορώ να πω πολύ συγκεκριμένα, γιατί γνωρίζω ε, καλά την πραγματικότητα στην πατρίδα μου, ότι οι γυναίκες ε, δεν διεκδικούν τόσο πολύ τα δικαιώματά τους, διότι μέσα στην οικογένεια είναι εκείνες που φέρουν το κύριο βάρος, δυστυχώς. δυστυχώς. Τώρα λοιπόν Έχουμε τις περικοπές, έχουμε την κρίση, έχουμε χαλάρωση των συνθήκων εργασίας, δηλαδή του ωραρίου εργασίας. Μπορεί να κληθεί ο εργαζόμενος να εργαστεί περισσότερες ώρες και ένα ημέρα, αλλά και αν εβδομάδα, πράγμα το οποίο δυσκολεύει πολύ τη δουλειά των γυναικών, γιατί έχουν πιο πολλή δουλειά ε, έξω από το σπίτι, αλλά η δουλειά στο σπίτι δεν μειώνεται. Πρόκειται λοιπόν για επίκαιρα προβλήματα. Πρόκειται για προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να εξετάσουμε ε, ανεξάρτητα από το ε, υπόλοιπο πλέγμα σχέσεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούμπερ για να απαντήσει. Δεν έχω συγκεκριμένες ε, πληροφορίες για το τι, πληρο... τι προβλέπει ο προϋπολογισμός για την προσέγγιση των φύλων. Δεν θα με εξέπλητε να γινόταν λόγος και για μείωση για μειώσει. Φαντάζομαι ότι περισσότερο θα πάμε προ την ευελιξία δεδομένων των πολιτικών προτεραιοτήτων και σε ένα χρονικό, σε ένα πλαίσιο μάλλον, σε δεδομένα όπου και η μετανάστευση και το άσυλο μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, τα πολιτικά δεδομένα. είναι ένα πρόβλημα στο οποίο το επενδύσουμε τόσο πολύ καιρό, που θα πρέπει επιτέλους να επιληθεί. Θα ήθελα ε, να υπογραμμίσω την ανάγκη να αναλυφθεί δράση, ώστε τα θέματα της ισότητας να ε, συζητηθούν. τα θέματα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθούνται ως προς τη διάσταση των φύλων γιατί πολλά από τα δικαιώματα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή και πρέπει οπωσδήποτε να επαχρυπνούμε. Όπως είπε η κυρία Ζούμπερ. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια μείζωνα αναμετατροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομική κρίση ανατρέπει πολλά πράγματα. Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι στο πολιτισμό οικονομικό πλαίσιο όλη η προσοχή δίνεται στις υποδομές και τις δομές ε, στη φροντίδα και τη μέρινα δεν υπάρχει. Πρόσβαση στη ε, μέρινα δεν αναφέρεται. Εάν ε, μπορούμε να διδαχθούμε από την κρίση του 2008, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αντιστάθμιση, αντίδραση στο, στην κρίση των ε, κρατικών χρεών και παράλληλη ανταπόκριση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίσει την ανάγκη για μια γενικότερη προσέγγιση που θα επιτρέπει στις γυναίκες να ασκούν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρούμπερι. Περνούμε στην κυρία Σιμονάτση, την επόμενη ομιλήτρια. Εξωτερικέ σχέσει. Έχετε κι εσείς 15 λεπτά στη διάθεσή σας. Για να μας παρουσιάσετε τα αποτελέσματα και την ανάλυση. εξωτερικές σχέσεις. Αντίθετα με τις άλλες παρουσιάσεις, μπορώ να πω ότι στις εξωτερικές σχέσεις βλέπουμε τη διάσταση του φίλου. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω πόσο σημαντικές είναι οι εξωτερικές σχέσεις ή διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική ενσωμάτωση, για την ανάπτυξη, για την ε, συνεργασία και διεθνή βοήθεια. Αυτή λοιπόν η διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική για την αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν έγγραφα στρατηγικής λοιπόν ε, δικής πολιτικής που υπογραμμίζουν τα, κύρια μέσα των ε, ευρωπαϊκών εξωτερικών δράσεων και που αναγνωρίζουν τη σημασία της ισότητας των φύλων και των σχετικών αρχών. Αλλά εδώ τέλειων ε, οι διαφορές, λέει η ομιλητρία. Διότι και πάλι στη συνέχεια ακολουθούμε την πορεία των άλλων εισηγήσεων. Ότι δηλαδή δεν εντοπίζονται σαφείς και δεσμευτικοί στόχοι ανάλογα με το φύλλο. Κύριες δράσεις, ορόσημα ορίζονται σε σχέση με πολιτικές αναφύλλου όπως η στρατηγική για την ισότητα μεταξύ και γυναικών 2010-2015 και το πρόγραμμα δράσης για τις γυναίκες στην ανάπτυξη 2010. Πλην όμως δεν έχουμε ενδείξεις ως προς το επίπεδο συμμόρφωσης και το συσχετισμό με τους στόχους. Το νομοθετικό πακέτο, η νομοθετική δέσμη μέτρων για την παγκόσμια Ευρώπη, όπως ονομάζεται αυτή η δράση, λέει τα εξή. Το Δεκέμβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νομοθετικό πακέτο ως τμήμα των προτάσεων για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο παρτιζόταν από μια κοινή ανακοίνωση ε, με στόχο Παγκόσμια Ευρώπη, μια, ένα κοινό κανονισμό για εξωτερικά μέσα και νομοθετικές προτάσεις για εννέα γεωγραφικά και θεματικά μέσα. Άλλα σημαντικά μέσα όπως η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική προστασία δεν περιλαμβάνονται μεν στο ε, πακέτο μέτρων αλλά θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται υπό το τίτλο Παγκόσμια Ευρώπη στην, στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να σας ε, δείξω τα κύρια δημοσιονομικά μέσα της ε, παγκόσμιας Ευρώπης. Στον τίτλο 4, Παγκόσμια Ευρώπη, έχουμε ως εξής τις συνολικές πιστώσεις για τα κύρια δημοσιονομικά μέσα. Κάποια μικρότερη σημασία τα έχω παραλείψει. Συνολικά έχουμε 70 εκατομμύρια ευρώ. 6,8% περίπου του όλου προϋπολογισμού. Μικρό σχετικά κεφάλαιο, αλλά πολύ σημαντικό πιστεύω για τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύρια θέματα λοιπόν μέσω αναπτυξιακής συνεργασίας, DCI, το πιο σημαντικό προς τους πόρους του, προενταξιακό μέσο, είπα, και μέσω Ευρωπαϊκής Γειτονίας, ΕΝΗ, Δεν θα τα αναφέρω όλα λεπτομερώ πριν, όμω ήθελα να επισημάνω ότι εδώ προβλέπεται ένα ακόμη δημοσιονομικό μέσο πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως, το οποίο όμως δεν υπάγεται στον προϋπολογισμό αυτόν. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει να ε, προσφέρει 34 εκατομμύρια ευρώ. Τι έχουμε κάνει λοιπόν. Από την ανάλυση των δεδομένων προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους κύριους στόχους α, ε, αναφύλο και ε, οι οποίοι καθοδηγούν τις διεθνείς και ανατομέα σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλύσουμε ποιοι από αυτούς τους στόχους μπορούν να ε, ικανοποιηθούν από τα υφιστάμενα δημοσιονομικά μέσα. Και προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε την εξής κατανομή. Στόχοι, ανα, στόχοι για τα φύλλα τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση, ένας από τους στόχους άλλωστε το η χιλιετίας. Βελτίωση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, της ε, υγείας των γυναικών, της πολιτικής ε, χειραφέτησης των γυναικών και τη θέση των πολιτών. Ε, πέρα της βίας που στηρίζεται στο φύλλο, υποστήριξη της ε, νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ε, μεταφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εάν προσέξετε θα δείτε ότι υπάρχουν δύο κυρίως μέσα, το μέσο για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία και για την ευρωπαϊκή γειτονία, τα οποία αντιμετωπίζουν τους πρώτους στόχους ιδιαίτερος. Πέντε προγράμματα λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτά, πέντε προγράμματα εντοπίζουν ε, το φύλλο σε έναν από τους τομείς τους οποίους ε, μπορούν να χρηματοδοτηθούν πράξεις υποστήριξης και κυρίως στο ε, τομέα της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Επιπλέον, εντοπίζουν ως θεμελιώδη, ως λόγο χρηματοδότηση μάλλον των δράσεών τους, την ισότητα μεταξύ των φύλων και έτσι αναγνωρίζουν και την οριζόντια φύση της υποστήριξης του στόχου της ισότητας των φύλων. Φερρυπίν, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας που είναι και το πιο ε, πλούσιο, με την καλύτερη πρικοδότηση, αναφέρεται σε δύο κύρια στοιχεία. Υπάρχει ένα γεωγραφικό πρόγραμμα δηλαδή, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της ε, τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας ε, μεταξύ των, ε, με τα τρίτα κράτη και υπάρχουν και δύο προγράμματα δράσεως προς όφελος όλων των απτυσσιωμένων ε, κρατών. Αυτά λοιπόν τα θεματολογικά προγράμματα απαντούν σε... στην ιδέα των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και την ε, στη συνεργασία με τι τοπικέ αρχέ αφετέρου. Εάν πάρουμε όμω την πρώτη κατηγορία, δηλαδή τα παγκόσμια δημόσια αγαθά, πρώτη κατηγορία, υπάρχουν πέντε μακροχώροι ε, χώροι οι τομεί μέσα σε αυτό το στο μεγάλο κεφάλαιο, που είναι το, το περιβάλλον και οι κλιματικέ αλλαγέ, η ενέργεια, η ανάπτυξη του ανθρώπου, η ασφάλεια των ε, τροφίμων, η, της προμήθειας τροφίμων και η μετανάστευση. Θέματα φύλου, διάσταση φύλου βλέπει κανείς μόνο στην, στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπου. Και όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα από την κυρία Ρούμπερη, είναι παράδοξο το ότι ζητήματα όπως η μετανάστευση δεν αναφέρονται στην, ε, με τη μέσα στη διάσταση του φύλου. Για να δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Στο μέσο γειτονία. Το μέσο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει την ε, δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρχές ισότητας, κράτους δικαίου, χρηστής διοίκησης και ανθρώπινης ανάπτυξης. Και εδώ λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφέστερη προσέγγιση με βάση τα φύλλα, χωρίς διακρίσεις για όλες τις δράσεις του κανονισμού. Όμως, παρά τη γενική υποστήριξη στην αρχή της ισότητας, το μέσο αυτό δεν προβλέπει συγκεκριμένους στόχους ή τομείς όπου, που να στοχεύει στην ισότητα των φύλων. Αντίστοιχα, ε, σχόλια μπορούσα να κάνω και για τα λοιπά μέσα, δεν έχω τον χρόνο όμως, μπορείτε να τα διαβάσετε στις ε, διαφάνειες, στα αντίγραφα. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αναφέρεται η διάσταση του φύλου, αλλά δεν υπάρχουν στόχοι και συγκεκριμένες δράσεις. Oh, yeah. Okay. So, eh, when we look at all these... Έτσι λοιπόν, όταν κοιτάμε όλα αυτά τα στοιχεία, προβλέπονται, αναφέρονται, ακόμη και συγκεκριμένες δράσεις προβλέπονται ορισμένες φορές, σε παραδείγματι στην περίπτωση των γεωγραφικών μέσων, βλέπουμε αναφορά Φερρυπίν μαζί με την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική ενσωμάτωση στη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, ως στόχος της ισότητας των φίλων, τη χειραφέτησης των γυναικών, θα πρέπει να επιδιώκεται. Αναφέρεται αυτό, αλλά χρηματοδότηση ή ειδικό δείκτης δεν αναφέρεται. Το ίδιο και για την Νότια Αφρική βία λόγω του φίλου η γενετήσια βία, το πρόβλημα του AIDS HIV, τομείς για τους οποίους λέμε ότι πρέπει να δοθεί χρηματοδότηση από το μέσο, αλλά χωρίς και πάλι συγκεκριμένες ενδείξεις. Νομίζω ότι τα τελευταία δεν θέλω να πω. Ένα μέσον το οποίο δεν έχει καμία αναφορά στα, στα φύλλα είναι αυτό που ονομάζεται μέσω, συνεργα... Ε, μέσω σχέσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αντιληφθούμε τι, ε, πώς μπορεί να γίνει ουδέτερος προς το φύλλο ένα μέσον. Το, με, το μέσο εταιρική σχέση, παραδείγματι, προβλέπεται ως ένα νέο μέσον για την ε, εξασφάλιση συνεργασίας για τρίτες χώρες που πλέον δεν δικαιούνται την αναπτυξιακή συνεργασία. Φερρυπίν, Αργεντίνη. Αργεντινή. Έχουν δηλαδή οι χώρες αυτές ε, ξεπεράσει το στάδιο της ε, μη ανεπτυγμένης χώρας, δεν έχουν φτάσει όμως στο επίπεδο της 100% ε, ανεπτυγμένης, αλλά δεν δικαιούνται την αναπτυξιακή βοήθεια. Τι προβλέπει, τι προσφέρει το ε, μέσο εταιρική σχέση. Προσφέρει οικονομικέ εμπορικέ σχέσει. Και είναι χαρακτηριστικό νομίζω το ότι δεν, υπάρχει, δεν προβλέπεται η ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φίλου μέσα σε αυτή την μορφή χρηματοδότηση της εμπορική ή της ε, οικονομικής σχέση. Δηλαδή θεωρείται ότι τέτοιου τύπου σχέσεις δεν χρειάζονται διάσταση φύλου. Αυτά τα έχω καλύψει λοιπόν εδώ. Μπορώ να προχωρήσω. Και θα ήθελα να απευθύνω μια προειδοποίηση ότι δεν είναι δυνατόν στο στάδιο αυτό του προγραμματικού κύκλου του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου να προσφέρουμε εκτίμηση ως προς τα κονδύλια που ενδεχομένως να αποδοθούν, να κατανεμηθούν μέσω των διαφόρων μέσων στον στόχο της σώτας των φύλων ε, πολλό δε μάλλον στην εξασφάλιση συγκεκριμένων στόχων ε, στις εξωτερικές δράσεις που εντοπίζονται για τα φύλλα. Όχι μόνο γιατί δεν ε, υπάρχει εγγραφή συγκεκριμένη για το φύλλο στον προπολογισμό αυτών κονδυλίων, αλλά και γιατί δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεδομένων σε σχέση με τους στόχους της ισότητας των φύλων από τα ισχύοντα μέσα εξωτερικής δράσης και ως προς την αξιολόγηση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας που αποτελεί και το κύριο εμπόδιο για την αξιολόγηση της επίπτωσης στο ε, στα φύλλα μάλλον των μέσων του μελλοντικού πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Επομένω, εφόσον δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε προηγούμενα προγράμματα, εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε μεσοπρόθεσμη ανάλυση των τρεχόντων προγραμμάτων, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα προσφέρει η επιπλέον χρηματοδότηση στην, ε, στα προγράμματα αυτά εξωτερική δράση σε σχέση με το φύλλο. Είναι ασαφή τα δεδομένα του παρελθόντο και δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε δηλαδή για να εκτιμήσουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Αναφέρθηκε και νωρίτερα από τον καθηγητή Βετίο, την καθηγήτρια Βετίο, ότι υπήρξε μια αξιολόγηση, μια απόπειρα αξιολόγησης, της, ε, του αντικτύπου, ε, της συνάφειας καλύτερα, των μέτρων αυτών ως προς το φύλλο και όσα έχει προτείνει ένα δίκτυ τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσω αυτού του συστήματος ε, καταγραφής απαιτείται για να συμπιληθούν να δίνουν τα κράτη-μέλη συγκεκριμένα απαντήσεις ως προς τα κονδύλια που λαμβάνουν από την ε, εξωτερική συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό. Καταρχάς πρέπει να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί ως προς την ερμηνεία που θα δώσουμε στα δεδομένα αυτά, διότι δεν ε, ελέγχονται, δεν εποπτεύονται όλα τα κράτη και όχι όλα τα κονδύλια. Φερρυπίν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά καλά αποτελέσματα, καλές επιδόσεις προς την ε, επιτήρηση αυτών των κονδυλίων. 88% των ευρωπαϊκών κονδυλίων υφίστανται αυτή την εποπτεία σε σχέση με την ε, λίστα του φίλου και συνολικά από τον ΩΣΑ 63,8%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν καταβάλει από ό,τι φαίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια στην ε, εποπτεία αυτή, στην επιθεώρηση των ε, κονδυλίων συνεργασίας με εστίαση στο φύλλο. Αλλά, εάν προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε τι είδους ποσοστά από τα ποσά αυτά απευθύνονται σε συγκεκριμένο φύλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο το 13% κατά μέσο όρο. όλων των ελεγχθέντων ποσών. 19,8% των ποσών είναι εστιασμένα από αυτά τα οποία ελέγχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για τον ΩΣΑ το ποσοστό αυτό είναι 33%. Αν κοιτάξουμε τώρα συγκεκριμένα τους τομείς, η εκπαίδευση και η υγεία είναι όντως, όντως θα, είναι οι πιο σημαντικοί τομείς η γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου βρίσκονται πολύ χαμηλά στον πίνακα συνάφειας ως προς την εστίαση στο φύλλο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ίσως θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερη προσοχή στα κριτήρια για την επαλήθευση και την αξιολόγηση. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω σύντομα στα συμπεράσματα τα μέσα των εξωτερικών σχέσεων που θα χρηματοδοτεί ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να έχουν θετική πλην όμως ε, μάλλον έμεση συνέπεια, έμεσο αντίκτυπο στους στόχους ισότητας των φύλων και αχειραφέτηση των γυναικών ή πρόσδοση δυνατοτήτων στις γυναίκες που εντοπίζονται από τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές ορίζουν τις εξωτερικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν μια σαφής στρατηγική αναφύλων ε, για στόχους, για ε, αναδια... ανακατανομή των ποσών δεν προκύπτει ως προς την κατάσταση εξωτερικές δράσεις που έχουμε αναλύσει και δεν μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τους πόρους που θα χρειαστούν για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί για, το, ε, για τα φύλλα. Η ισότητα των φύλων θεωρείται μια βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προάγεται και να ενσωματώνεται σε όλα τα διαφορετικά στάδια του προγραμματισμού των εξωτερικών δράσεων και, στη, και έχει τεράστια σημασία για την καταπολέμηση της φτώχειας, κύριο στόχο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ε, παρεμβάσεις ως προς την ε, ισότητα των φύλων και η ανακατανομή των ποσών θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το πόσο είναι ενσωματωμένη σε ε, στρατηγικές ανακράτωση περιφέρεια και τα πολιετή ε, σχέδια ίδια σας του φύλου. Αναφέρθηκε και νωρίτερα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια αξιολόγηση εκ των προτέρων, αλλά και επίσης αξιολόγηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Μια τελευταία, μια τελευταία παρατήρηση, μια και έχω ξεδλήσει το χρόνο μου. Αναφέρθηκε νωρίτερα ότι η ενσωμάτωση της τάσης των φύλων, τα φύλλα γενικά είναι, ε, κινδυνεύουν να γίνουν αόρατα στη στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σε εξωτερικές σχέσεις έχουμε την, τον αντίθετο κίνδυνο, ε, δηλαδή ότι μπορεί παντού να αναφέρεται η διάσταση των φύλων, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες δράσεις και χρηματοδότηση και αυτό νομίζω είναι το ο πιο ε, σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε στι εξωτερικές μα σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σχόλια, ερωτήσει υπάρχουν. Παρακαλώ. Είμαι πολιτικός σύμβουλος της ομάδας των Πρασίνων αναφορικά με το ζήτημα του δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Για να πω το εξής. Από την αρχή κάνετε ένα διαχωρισμό των μέσων στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου και κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν μελέτες ή στοιχεία τα οποία δείχνουν κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης έχει ε, επιπτώσεις ε, σε θέματα ισότητας ε, φύλων, διότι τα χρηματοδοτικά μέσα της εξωτερική πολιτική βρίσκονται μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και υπάρχει έλεγχο του Κοινοβουλίου και το ταμείο, το Αναπτυξιακό Ταμείο βρίσκεται εκτό. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το Αναπτυξιακό Ταμείο αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα ή όχι και αν είναι λιγότερο καλά τα αποτελέσματα από ό,τι πιστεύω ότι δεν έχω στοιχεία θα ήταν ένα πλέον επιχείρημα έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο μέσα από το δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό προ όφελο των γυναικών. Η κυρία Σιμονάτση έχει το λόγο. Ναι, ε, υπάρχει μελέτη του Ταμείου ανάπτυξη Δεν ήταν μια σε πάθος μελέτη και ανάλυση, αλλά μπορούμε να πούμε πως ε, υπάρχουν τα ίδια προβλήματα σε ό,τι φορά την στόχευση αλλά και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των προγραμμάτων. Το γενικότερο σχόλιο λοιπόν της ανάγκης ε, παρακολούθησης, ε, αξιολόγησης σε κάθε φάση αλλά και στο τελικό στάδιο των ταμείων θα ε, εφαρμόζεται και στο ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα συνάγω λοιπόν κάποια συμπεράσματα και ως εκ τούτου θα μιλήσω την Σουηδική φορές τα ακουστικά σας. Να ευχαριστήσω όλους και όλες τους εμπειρογνώμονες. Ήταν πολύ σημαντικά τα όσα ακούστηκαν σήμερα εδώ. Είναι ζητήματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα ξεχάσουμε ότι δηλαδή η διάσταση του φίλου θα πρέπει να είναι πανταχού παρούσα. Πολλά από αυτά θα μας χρησιμεύσουν κατά τον των εργασιών μας. Κυρία Μπέτιο. Αναφέρθηκε στους, στα εισοδήματα των γυναικών, των ανδρών και αυτό το χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στα εισοδήματα αλλά και μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολύ δρόμο ε, να διανύσουμε για να πετύχουμε την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Επίσης ε, πολλά έχουμε να κάνουμε για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο του 75%. Ναι, το ζήτημα είναι να μην έχουμε μόνο στόχους, αλλά έχουμε και τους κατάλληλους δείκτες, κυρία Μιλντέρμα, Εβεβαιώσατε αυτή την έλλειψη ισορροπίας που διαπιστώνουμε. στο θέμα της ε, Εκπαίδευση αλλά και ειδικά σε ό,τι φορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ισότητα των φίλων λοιπόν και η διάσταση αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε όλους του. τομείς. Κυρία Λιμπεράκη, επίσης ε, μιλήσατε για το ζήτημα της υγείας και ιδιαίτερα των ε, προσώπων αν των 50 και ότι σε όλα τα κράτη-μέλη ε, γυναίκες που πάσχουν από χρόνες ασθένειες άνω των 50 είναι περισσότερες σημαντικά από τους άνδρες μόλον ότι ζουν περισσότερο ε, επίση στο δείκτης της ε, ευτυχίας ήταν και αυτό ένα ενδιαφέρον θέμα. οι στόχοι οι γενικοί που περιλαμβάνονται σε στρατηγικά έγγραφα, έγγραφα πολιτικής ε, σε πολλούς ε, τομείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να συμπεριλάβουν την διάσταση του φίλου Του φίλου. Αλλά παράλληλα όπως είπαμε χρειάζεται να έχουμε και τους κατάλληλους δείκτους, δείκτες για να τα υπολογίσουμε. σημασία έχει να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε στατιστικές αναφύλο. Διαφορετικά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα. Και τέλος η κυρία Σιμονέτση ε, μίλησε για μια σειρά από ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα Ε, ήταν όλα ενδιαφέροντα ε, αυτά που μας είπε, διότι έθιξε επίσης και το ζήτημα της ε, γεωργίας, ε, επίσης το ζήτημα των μεταφορών. Η μεταφορά είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Και αν δεν υπάρχει εδώ η συμπεριληπτιάσταση των φίλων, αυτό μπορεί να αποβεί εις βάρος των γυναικών και της δυνατότητας ε, μετακίνησής τους. Μας δώσατε λοιπόν πολλά όπλα για να χρησιμοποιήσουμε στο οπλοστάσιό μας, ε, πολλά βέλη για την φαρέτρα μας και που, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και το κοινό.